Colleghi, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μια φορτωμένη ημέρα μπροστά μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινήσουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού σχετικά με τη διαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Κωσυφοπεδίου. Εισηγητής ε, η συγγήτρια μάλλον η κυρία Λούνα Τσεκ βρίσκεται εδώ εντός της αιθούσης. Bene, compromesso 1. Συμβαστική τροπολογία υπαρθμών 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφικά κατά δεκτό δεύτερο τμήμα ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και το δεύτερο τμήμα υπαριθμών συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2 ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία υπερθυμών 48, ψηφιπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Υπερθυμών 49, ψηφιπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπερθυμών 3, ψηφιπέρ, κατά αποχές δεκτή. Υπαριθμόν 60 τροπολογία με προφορική τροπολογία του εισηγήτριας. Διαγράφονται οι λέξεις with satisfaction με ικανοποίηση ψηφίζουμε ψηφί πέρα κατά δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 4 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εβδομήντα τέσσερα ψήφι κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 5 ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπερθμό 86 ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 88 ψήφι υπέρ. Κατά. εποχές... Δεκτή. Συμβαστική υπερθυμών 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπερθυμών 100. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία σε αυτήν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Υπάρχει 101 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. 102 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε επαλήθευση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός. Αποτέλεσμα ψηφοφορίας 33 ψήφοι υπέρ, 18 ψήφοι κατά. Δεκτή η τροπολογία. Υπερθμόν 7 συμβαστική υπέρ. Με διορθώνουν. Πρέπει να ψηφίσουμε η τροπολογία 103. Ψήφι υπέρ της 103. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 104 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 112 με προφορική τροποποίηση της εισηγήτριας. ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 με χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ ψήφι κατά αποχές δεκτή, δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 με προφορική τροπολογία της εγκύρια ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 125. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Φαίνεται πως απορρίφθηκε, αλλά ε, δεν ψηφίσατε όλοι. Παρακαλώ, ας επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της 125. απορρίπτεται με δύο ψήφους, μάλλον με μία ψήφο. Η συνάδελφος δεν ψήφισε, παρατηρεί η συγκεντρία. Άρα πρέπει να καταμετρήσετε την ψήφο υπέρ. Συν τη δική μου ψήφο υπέρ. Ούτως ή άλλως απορρίπτεται με ισοψηφία. Πάντα με ευχαρίστηση ακούμε τη φωνή σας. 124. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση με αναγκάζεται παρακαλώ να ψηφίσετε επί της 128 Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Περνάμε στην 130. Περ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 131. Λοιπόν, μου ζητάνε ηλεκτρονική επαλήθευση. Επανερχόμεθα στην 130. Παρακαλώ, ψηφίσατε ηλεκτρονικός επί της 130. Συγγνώμη, δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου, Πρόεδρο. Εντάξει, πείτε μας τι ψηφίσετε, υπέρ. Ωραία. Άρα συν δύο ψήφοι υπέρ Λούνατσεκ και εσείς ολοκληρώνετε η ψηφοφορία. 35 ψήφοι υπέρ, 20, 37 ψήφοι υπέρ, συγγνώμη, 23 κατά. Περνάμε στην 131. Εκατόν τριάντα ένα επαναλαμβάνω. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή Περνάμε στην 144 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 100 152 ψήφι υπέρ 152 κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 155. 156. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Συμβαστική 12 ψη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 172 ψήφι κατά. Ας ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφορία. Εντάξει. Οι γνωστοί δύο ψήφοι υπέρ. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 173. Έγινε δεκτή 172 φυσικά. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 173. 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή 176 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία συμβαστική υπαριθμό 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 181. Τροπολογία 181 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Με 182 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Με 183 υπέρ κατά αποχές δεκτή 185 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 186 υπέρ κατά αποχές δεκτό 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 188 υπέρ κατά αποχές δεκτό 189 υπέρ κατά αποχές δεν ψηφίσατε όλοι, ας επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός ε, Τροπολογία 189. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε διότι υπάρχουν δύο επιπλέον ψήφοι κατά. Απορρίπτεται λοιπόν η τροπολογία 189, 190, 191. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να είναι προφανή, ήταν προφανές το αποτέλεσμα. Περνάμε στην 192 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 193 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 194 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 195 υπέρ κατά αποχές δεκτή 197 96 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία 197 Μητροπολία 197 ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 198 υπέρ κατά αποχές δεκτή 199 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε τροπολογία 199 Κοιτάξτε, υπάρχει ένα συνάδελφο τη σοσιαλιστικής ομάδας επιπλέον, υπεράριθμος, δηλαδή ψηφίζει δίχω να έχει το δικαίωμα. Ο Παντσέρη λέει πως οι σοσιαλιστές ποτέ δεν περισσεύουν, αλλά κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Αποτέλεσμα, έγινε δεκτή η τροπολογία 199 Καλωσορίζουμε τον ε, πραγματικό πρόεδρο της Επιτροπής. Ε, Καλώς Χέλμουντ ε, Χέλμουτ Μπρόκ. Και χρόνια πολλά. Έχετε τα σου. Τροπολογία 200. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται 202 ε, υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 204 Έχει ζητήθει χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου. Περνάμε στην τροπολογία 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά αποχές Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Λίγοι ψηφίσατε και άρα είναι δύσκολο να καταλάβουμε την βούληση της Επιτροπής. Μα η βούληση έγκυται στην καρδιά, Πρόεδρε. Δεν εκδηλώνεται πάντα. Ολοκληρώθηκε η τροπολογία, εγκρίθηκε η, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, εγκρίθηκε η τροπολογία, συγγνώμη. Με συντριπτική πλειοψηφία. Μίλησε η καρδιά. Τροπολογία υπερθμών 2. Υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Περθμόν 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Εποχές ε, δεκτή. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 10. Χρειάζεται λίγο χρόνο για να λειτουργήσει το μηχάνημα. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή η τροπολογία 10. 39 υπέρ, 23 ψήφι κατά. Τροπολογία 11 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. <clears throat> κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 13 ψήφι Κατά αποχές δεκτή τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Υπέρθυμο 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά Λίγοι ψηφίζετε, δεν ξέρω τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός. Τροπολογία 16, παρακαλώ, ψηφίσατε ηλεκτρονικός. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε, 43-15, τροπολο... τροπολογία 1, υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. <clears throat> Και το τελική ψηφοφορία επί του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Έληξη ψηφοφορία. Συντηρητική πλειοψηφία υπέρ. Συγχαρητήρια κυρία Λούνατσοκ 54. 6 το αποτέλεσμα. Va bene, passiamo la vuole chiarire una cosa un attimo. C'è la richiesta di, di interrompere per 5 minuti. Υπάρχει αίτημα για διακοπή της συνεδρίασης επί 5 λεπτού προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συναδέλφων. Παρακαλώ 3-5 λεπτά διάλειμμα, αναμονή. Mm, va bene.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

If adesso. Colleghi, colleghi, riprendiamo i lavori. Επαναλαμβάνουμε τις εργασίες μας, συνάδελφοι. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ Συνάδελφε Ουλουρίκε, καθίστε. Θα ψηφίσουμε την έκθεση πρόοδου του 2004 για την πρώην Ιουγκουλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ξεκινάμε με την τροπολογία παρθμών 1, είναι προφορική τροπολογία, ψηφίπερ Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 3 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 41 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 45. Υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Ελάχιστοι συνάδελφοι ψήφισαν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 45, ηλεκτρονικός, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της μεγάλη η υπερπλειοψηφία, τροπολογία 46. Έχουμε την προφορική τροπολογία του υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, εποχές, δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, εποχές δεκτή. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Ο. Διαμαρτυρίες από την αίθουσα. Εντάξει, α, εφόσον το επιθυμεί η κυρία Λούνατσεκ, ε, θα περάσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της 57. το λέγει το όνομά της. Λούνα Τσεκ. Δεν έχουν ψηφίσει όλοι οι συνάδελφοι, παρακαλώ ψηφίσατε. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία απορρίπτεται. Τροπολογία 66 Υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται 67 Υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται 68 Υπέρ κατά εποχές ας επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία έληξε η ψηφοφορία εγκρίνεται τροπολογία 69 Τροπολογία 69 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 70. Ε, κοιτάξτε, ήταν, είναι προφανές ε, εγκρίθηκε. 70 υπέρ. Κατά. Εδώ σε επαληθεύσουμε καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 70. Έληξε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 71. Ο κύριος Κούκεν ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια προφορική τροπολογία επί της 71 να διαγραφεί η λέξη διαιτησία, μηχανισμός μεσολάβησης και ε, από μεσολάβηση να γίνει διατησία. Η υπόλοιπη παράγραφος με έχει. Ευχαριστώ. Συμφωνείτε με την προφορική αυτή τροπολογία. Όχι. Υπάρχει κάποιος ε, που διαφωνεί. Άρα θα περάσουμε στην ψήφιση του κειμένου ως έχει. Ψηφίζουμε λοιπόν επί του τροπολογίας 71 ως έχει. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται 76 όχι, όχι, συγγνώμη καταπίπτει εφόσον εγκρίθηκε η συμβαστική τροπολογία υπερθυμών 7 περνάμε στην τροπολογία 81 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 Θέλετε να επαληθεύσουμε την 81, ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικό επί του 82, άρχεται ψηφοφορία. Ακόμα τρεις να απομένουν να ψηφίσουν. Πέρα ψηφοφορία. εγκρίθηκε η τροπολογία. Περνάμε στην 83. Ψήφι Κατά Αποχές εγκρίθηκε. 85. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Προφορική τροπολογία υπερθυμών 3 του συναδέλφου Κούκαν υπέρ κατά αποχές δεκτή. 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ <clears throat> παρατηρήσεις του μικροφόνου Δεν θα έπρεπε να την διαβάσετε. Όχι, όχι, όχι. Δεν χρειάζεται, συγγνώμη. Τροπολογία 108. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 109. Όχι, όχι, όχι. Περνάμε στην τροπολογία 12 τη συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβεστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 με την προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ αποχές κατά δεκτή 124 129 συγγνώμη ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 136 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 139 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 142. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε. 142. Τροπολογία. Έχουμε τέσσερις συνάδελφοι απομένουν. Έληξε η ψηφοφορία, έγινε δεκτό το πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα της 142, ψήφι περ, κατά, αποχές, απορριπτέται. 143 με προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 όχι καταπίπτει καταπίπτει 145 συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 104 τροπολογία υπέρ. Κατά. Πολύ λίγοι ψήφισαν, ας επαληθεύσουμε. 104. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστη της ψηφοφορίες. μεταπεινώνεται. Η καρδιά μιλάει, πρόεδρε, η καρδιά μιλάει. Τροπολογία, ε, συμβαστική 19, συγγνώμη. Συμβαστική 19, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. Τροπολογία 150, υπέρ κατά αποχές δεκτή 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154. Ζητήθηκε επαλήθευση για την 153 του Αντιπρόεδρου κ. Κόβατσεφ. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικός. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφων, αλλά απορρίφθηκε 154 υπέρ κατά αποχές να εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία, η κυρία Γιαννάκου ζήτησε το λόγο. Πρόεδρε, στην τέταρτη γραμμή, στο συμβιβασμό 20, λέει εκπαιδευτικά προγράμματα με τη Βουλγαρία, μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας. Αλλά δεν υπάρχει τροπολογία που να αναφέρει την Ελλάδα. Μόνο τη Βουλγαρία αναφέρουν. Γι' αυτό ζητάμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Δηλαδή πρώτα χωρίς τη λέξη Ελλάδα και αν απορριφθεί και με την Ελλάδα. Χωριστή ψηφοφορία. Όχι σε τμήματα, χωριστή. Χωριστή. σαφές το αίτημα της συναδέλφου, το λόγο ζήτησε ο συνέλφος Χόουιτ. Ναι, για αυτούς που δεν πήγανε στη συνεδρίαση για τους συμβιβασμούς. Εγώ και η Σκιώδης αποφασίσαμε να παραμείνουμε στην ορολογία που χρησιμοποίησε την προηγούμενη φορά το Κοινοβούλιο. Δέχομαι το αίτημα της κυρίας Γιαννάκου να γίνει χωριστά η ψηφοφορία, αλλά εγώ θα ζητήσω και σε αυτήν να διατηρήσουμε την προηγούμενη διατύπωση. Allora. Ok, allora votiamo, vi chiedo di votare. Λοιπόν, ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία 20 δίχως τον όρο Ελλάδα. Ελλάς. Ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτό. Και τώρα ψηφίζουμε με, την συμπερίληψη της, ε, του όρου Ελλάς. Ψήφι ψήφι κατά. Α, όχι, όχι για τη συμπερίληψη του όρου Ελλάς. Μα ψηφίσαμε την πρώτη φορά χωρίς τη λέξη Ελλάς και τώρα ψηφίσαμε μετά για την ίδια τροπολογία αλλά με την λέξη, με τη λέξη Ελλάς. Va bene, allora abbiamo votato sul... Κοιτάξτε, ψηφίσαμε επί του πρώτου αιτήματο ε, που προβλέπει στο συμβασμό 20 να μην συμπεριληφθεί ο όρος Ελλάς. Τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε για τη συμπερίληψη του όρου Ελλάς ε, στην τροπολογία 20, τη συμβαστική τροπολογία 20. Ε, Κατέστην σαφής, πρόκειται για μια χωριστή ψηφοφορία σε τμήματα. Ψηφίσαμε επί του πρώτου τμήματος λοιπόν και τώρα θα ψηφίσουμε επί του δεύτερου τμήματος της Συμβαστικής 20. Το πρώτο τμήμα αποκλείει τον όρο Ελλάς, το δεύτερο τμήμα τον συμπεριλαμβάνει. Αυτό μου λέει η γραμματεία και δεν έχω καμία αμφιβολία πως πρόκειται για την ορθή ερμηνεία. Ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για να μην υπάρχουν ενδεχόμενε αμφισβητήσεις. Σας ζητώ λοιπόν να ψηφίσετε τώρα σου σύμφωνα με τα όσα σας ζητήθηκαν. Για τη συμπερίληψη του όρου Ελλάς. Va bene? Allora vi Ωραία. Λοιπόν, ψηφίσατε ηλεκτρονικώς για την συμπερίληψη του όρου Ελλάς στην συμβαστική τροπολογία 20. Ακόμα τρεις συνάδελφοι απομένουν πέρα ψηφοφορίας και εγκρίθηκε λοιπόν η συμπερίληψη του όρου Ελλάς. Τροπολογία 159 ψήφι πέρα κατά απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 8. Η ζητή χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 8 υπέρ κατά αποχές ας επαληθέψουμε. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 8. Παρακαλώ ψηφίσατε ηλεκτρονικός. Πέρασε της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 14 για να ακούσω υπέρ Κατά. Εποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. τέσσερα, όχι, καταπίπτει, καταπίπτει, διότι έγινε δεκτή η 3. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός θα ψηφίσουμε. πέρα τη ψηφοφορία ε, με συντηρητική πλειοψηφία έγινε δεκτή. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Κάνουμε μια διακοπή για διαβουλεύσεις ε, σχετικά με την επόμενη ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στην ψήφιση τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η συγγήτρια κυρία Νέιτς, ηλεκτρονικός παρακαλώ ψηφίστε. Τέσσερις ακόμα συνάδελφοι από μένα ψηφίσουν, ε, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Συντριπτική πλειοψηφία. 59 υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια κυρία εισηγήτρια. Il vero interprete del popolo. Bene, Συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 14, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου ε, για το Μαυροβούνιο το 2011. Εισηγητή ο συνάδελφος Τάνοκ, ε, όπως γνωρίζετε το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις ε, με το Μαυροβούνιο ή μάλλον αποφάσισε ότι οι διαπραγματεύσεις ε, με το Μαυρομού θα πρέπει να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2012. Στην έκθεσή του, ο κ. Στάνο εξετάζει τι πολιτικέ επιπτώσει αυτή τη απόφαση και άλλε πτυχέ τη διαδικασία ένταξη ε, του Μαυροβούνιου. Κύριε Τάνοξ, σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ξανασυγχαίρω για την επανεκλογή σας εχθές. Εδώ πρόκειται για τη δεύτερη έκθεση που έχω την τιμή να παρουσιάζω στην Επιτροπή σας κατά την εντολή αυτή. Αφού είχα οριστεί μόνιμος, λέει, εισηγητής για αυτό το θέμα. Δεν είναι κανένας τίτλος πολύ τιμητικός, αλλά τέλο πάντων είναι η δεύτερη έκθεση μου από τότε που το Μαυροβούνιο έγινε επισήμως υποψήφια χώρα για ένταξη τον Δεκέμβριο του 10 και τώρα απολαμβάνει και την απελευθέρωση των θεωρήσεων και μετακίνηση μέσα στο χώρο Σέγγεν από το 9. Ακούστηκαν σχεδόν σουρεαλιστικά σχόλια εχθές για την ένταξη της Μακεδονίας. Φαντάζομαι τι θα πούνε και για τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και την Αλβανία. Το Μαυροβούνιο πάντως είναι απλή χώρα για εξέταση όσον αφορά τον μόνιμο εισηγητή σας τουλάχιστον, ιδιαίτερα ως προς το θέμα της αξιολόγησης της προόδου του προς την οδό της ένταξης. Επίσης πιστεύω ότι τα σχόλια του Επιτρόπου Ρέναν δεν απατώμε, είχε πει ότι η ένταξη του Μαυροβουνίου είναι <clears throat> κάτι απλό χωρίς προβλήματα και αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Τη τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου που ανέβαλε την αρχή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, κάτε με, το σχόλιο αυτό ήταν απογοητευτικό για τη χώρα και για την ηγεσία της και νομίζω ότι η απόφαση αυτή τα βασιζόταν σε πολιτικά και εσωτερικά κριτήρια μάλλον παρά σε αντικειμενικά και οφειλόταν και στη γενικότερη αντίληψη που έχει τώρα η Ένωση για τις προσεχείς διευρύνσεις και δεν αφορούσε μάλλον την ε, πρόοδο που έχει κάνει το Μαυροβούνιο για την επίτευξη των στόχων και κριτηρίων που του έχουν τεθεί. Θα έλεγα μάλιστα ότι κατ' εμένα το Μαυροβούνιο δεν δικαιολογεί καθόλου τις καθυστερήσεις αυτές. Οι τομείς που, όπου ζητήθηκαν βελτιώσεις, δηλαδή η εργασία του Κοινοβουλίου, οι γενικές του διαδικασίες, ο εκλογικός νόμος, η μεγαλύτερη επαγγελματικότητα στη διοίκηση, είναι βέβαια πολύ μικρή χώρα και έχει πολύ λίγους δημοσίου υπαλλήλους, η ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα, η καταπολέμηση της διαφθοράς και δωροδοκίας και του οργανωμένου εγκλήματος που είναι πρόβλημα ολόκληρης περιοχής, η ελευθεροτυπία και η ελευθερία του λόγου και οι κατηγορίες που ακούστηκαν για επιθέσεις ή πιέσεις κατά ορισμένων δημοσιογράφων ή εφημερίδων μεγαλύτερη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών για όλα αυτά στο ψήφισμά μου λέω Μιλάω για την οικονομία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τώρα το Μαυροβούνιο για την ανάπτυξή του. Δεν είναι βέβαια τμήμα της Ευρωζώνης αλλά χρησιμοποιεί ήδη το ευρώ. Παράδοξο θα φανεί σε μερικούς. Και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει οφείλονται και στη χρήση αυτού του ναμίσματος. Η κρίση και η ύφεση οι μεταρρυθμίσεις στι συντάξεις και η καταπολέμηση περικοπή της γραφειοκρατίας η αύξηση των ε, εξωτερικών επενδύσεων και η δημιουργία ενός καταλληλωτέρου επιχειρησιακού κλίματος ε, είναι θέματα που έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Μία-δύο χώρες βέβαια ίσκησαν βέτο για την ένταξη του Μαυροβουνίου στον ΠΟΕ και αυτό το λέω στην έκθεσή μου και συζητώ θέματα που αφορούν τα κύρια πολιτικά κριτήρια που αφορούν μια ένταξη στην Ένωση όπως διεθνωτικές σχέσεις. Βέβαια το Μαυροβούνιο είναι μικρή χώρα και με αρκετή εθνοτική ενότητα και το θέμα της χρήσης της σερβικής γλώσσης αντί της μαυροβουνικής είναι κάτι που δεν το αναφέρω πολύ γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Το θέμα της μεταχείρισης αναπήρων ή του δικαιώματος επιστροφής εκτοπισμένων και εξορίστων σε διάφορα τμήματα της πρώην Νοτιοσλαβίας. Ε, δεν έχει ακόμα λυθεί αλλά σημειώθηκε πρόοδο Το θέμα της ανεξαρτησίας του δικαστικού τομέα και της ελευθεροτυπίας δεν έχει προβλήματα ιδιαίτερα. Επίσης έθεσα θέματα εκλογικά και ενεργειακά. Το Μαυροβούνιο ευτυχώς έχει πολλούς υδροηλεκτρικούς πόρους για το περιβάλλον και τον τουρισμό το Μαυροβούνιο υπερηφανεύεται ότι είναι χώρα ε, πολύ ευαίσθητη στα περιβαλλοντολογικά. Έχει πολλές φυσικές καλονές ιδιαίτερα την σακτές του και άρα έχει και υψηλό τουρισμό. Τέλος, η περιφερειακή συνεργασία με τους γείτονές του υπάρχει μία μικρή συνοριακή διαφορά με την Κροατία και θα ξέρουν οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχει θέμα εκεί καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος. Υπάρχουν όμως διμερείς συνθήκες ε, μη έκδοσης ή έκδοσης μάλλον μεταξύ Μαυροβουνίου, Σερβίας και άλλων πρώην Ιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 2 Φεβρουαρίου και προσβλέπω με αδημονία στις, ε, στα σχόλια των ε, συναδέλφων πέρυσι η περσινή μου έκθεση ήταν από, πέρασε πολύ εύκολα χωρίς ούτε μία ψήφο κατά και πολύ λίγες τροπολογίες κατατέθηκαν. Ίσως φέτος κατατεθούν περισσότερες, θα το δούμε. Γενικά όμως νομίζω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να στηρίξει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο όσο το δυνατόν νωρίτερα. Νομίζω ότι το Συμβούλιο προβλέπει τον Ιούνιο, δεν ξέρω γιατί τον Ιούνιο, αλλά δεν θα τα σώμουν κατά. Ορίστε σας ευχαριστώ αυτά. Κοιτάξτε, στο σημείο αυτό ξεκινάει η συζήτηση με τους σκιώδεις ηγητές. Η συνέλφος Ιμπριζάτσιτς έχει το λόγο. Παρακαλώ να παραμείνετε εντός του τριλέπτου Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Τάνοκ και με την αξιολόγησή του για την πρόοδο του Μαυροβουνίου. Είναι από τις απλούστερες περιπτώσεις που χρειάστηκε να συζητήσουμε ποτέ για προενταξιακή αξιολόγηση. Και συμφωνώ επίσης με αυτά που είχε πει ο Όλι Ρεν και ο Επίτροπος Βούλε πιο πρόσφατα, ότι δηλαδή το Μαυροβούνιο είναι success story. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η περιφέρεια ως προς τη συνεργασία με γειτονικές χώρες και εντάσεις εσωτερικές, εθνοτικές, όλα αυτά τα προβλήματα δεν παρατηρούνται στο Μαυροβούνιο. Το κείμενο όπως μας το παρουσιάσανε σήμερα μου φαίνεται πλήρες και τα σημεία που θέλω να σχολιάσω ιδιαίτερα ε, δεν χρειάζονται τροπολογίες γιατί το κείμενο γενικά είναι καλό. Έχουμε ακόμη μερικές μέρες για να σκεφτούμε την κατάθεση τροπολογιών. Αν τελικά καταθέσω θα αφορούν ε, λεπτομέρειες διακοσμητικά θέματα καλοπιστικά καλοπισμού του κειμένου αλλά όχι αμφισβήτηση της ουσίας της έκθεσης ή θεμάτων άλλων ουσιαστικότερων γιατί τα κάλυψε όλα ο κύριος Τάνοκ οικονομία, πολιτική, συνεργασία με γειτονικέ χώρες απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην προηγούμενη δηλαδή έκθεση του Μαυροβουνίου λήφθηκαν αυτά υπόψη εκ νέου. Είναι σημαντικό να συνεχίσει λοιπόν το Μαυροβούνιο τις μεταρρυθμίσεις του και να αναγνωρίσουμε όλες τις προόδους που έχει κάνει. Αναμένω και εγώ να δω τα σχόλια των υπολείπων συναδέλφων και τις τροπολογίες τους. Βασικά όμως συμφωνώ με το κείμενο που μας παρουσίασε ο κύριος Τάνοκ. Ε? Ο Σνέλος το λόγο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τάνοκ, διότι η έκθεσή του βασικά είναι πολύ καλή. Και εγώ είμαι σκιώδης για τους σοσιαλιστές. Θα καταθέσουμε μερικές τροπολογίες, αλλά και πέρυσι είχε πει τα βασικά, απλώς το βελτίωσε αυτή τη φορά. Γενικά συμφωνούμε και θα συμφωνήσουν νομίζω και οι περισσότερες πολιτικές ομάδες γενικά για την κατάσταση στο Μαυροβούνιο. Παρόλα αυτά μπορεί να καταθέσουμε μία-δύο τροπολογίες αλλά δεν είναι πολύ βασικές σε δύο ή δύο τομείς που πρέπει να ξαναδούμε τη διατύπωση. Ένα για τη διαφυθορά και το, την ένωμη τάξη το κράτος δικαίου. Εδώ το Μαυροβούνιο έχει κάνει ίσως λίγο λιγότερη πρόοδο αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ασκήματα πράγματα γιατί το θέμα βέβαια δεν είναι πώς θα αλλάξουν οι κανόνες γραπτά, αλλά στην πράξη. Να αλλάξουν οι αξίες στην κοινωνία του Μαυροβουνίου. Μερικά σημεία θέλουμε να τα ενδυναμώσουμε και το ίδιο ισχύει και το δεύτερο τομέα, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών. Ο κύριος Τάνοκ μας μίλησε για την ισότητα των φύλων πολύ ωραία Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η κατάσταση της αγοράς εργασίας όπου θα μπορούσαμε να είμαστε σαφέστεροι. Και επίσης of, e πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση από την ΕΠΑ. E και συμφωνώ με τον κύριο Τάνοκ ότι δεν πρέπει το Μαυροβούνιο να καθυστερήσει στις διαπραγματεύσεις λόγω της κατάστασης που ισχύει σε άλλες χώρες των δυτικών λεγόμενων Βαλκανίων. Εθνικά συζητιέται πολύ το θέμα της διεύρυνσης και δυστυχώς οι ευρωπαϊκές χώρες συνήθως παρετούνται από τα αιτήματα των υποψηφίων χωρών για ένταξη. Αλλά κάθε θέμα πρέπει να συζητιέται από μόνο του, όχι μέσα σε σύνδεση με εσωτερικά προβλήματα. Το, αυτό ισχύει και για το Μοντενέγκρο, το οποίο έχει κάνει μεγαλύτερη πρόοδο από άλλες χώρες γειτονικέ. Μπορεί λοιπόν να καταθέσουμε μία-δύο τροπολογίες, επαναλαμβάνω, αλλά δεν θα είναι πολύ βασικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Βάιγκλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ για την φιλόδοξη και δημιουργική προσέγγιση που είχε στην έκθεση αυτή. Επίσης ε, τον ευχαριστώ για το ότι είναι σύντομη αυτή η έκθεση. Είναι ένα μικρό κράτος, ε, διάφανο θα έλεγε κανείς και νομίζω πως μπορούμε να δείξουμε μια θετική προσέγγιση όσον αφορά την πρόοδο του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να είμαστε σύντομοι. Δεν ε, υπάρχει λόγος να καταθέτουμε πολλές ε, τροπολογίες. Έχουμε λίγα μόνο σχόλια που νομίζω πως πρέπει να συμπεριληφθούν στο έγγραφο αυτό. Συμφωνώ και υποστηρίζω την ιδέα που μόλις εξέφρασε ο συνάδελφος των σοσιαλδημοκρατών. Δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσει η έναρξη των διαπραγματεύσεων και ελπίζω σε όλα τα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει συμφωνία πως το Μαυροβούνιο είναι επιτυχημένη περίπτωση, είναι θετικό παράδειγμα, δεν υπάρχουν προβλήματα στον ορίζοντα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα επίση να τονίσω πως το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει πρόοδο σε κάποιους κρίσιμους τομείς που αναφέρθηκαν, ειδικά αναφέρομαι στην ε, διαφθορά. Νομίζω είναι σωστό να λέμε πως το Μαυροβούνιο έχει κάνει συνειδητή προσπάθεια και έχει σημειώσει πρόοδο, έχει σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες και βεβαίως είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με την Ιντερπόλ. Το επόμενο θέμα τώρα, η ελευθερία των ΜΜΕ και τα περιστατικά που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα, έτη. επιθέσεις ε, σε δημοσιογράφους ε, που ήταν ε, θεωρούνταν πτέσματα, αν θέλετε, και ανάλογα αντιμετωπίζονταν. Εν πάση περιπτώσει τα περιστατικά αυτά έχουν μειωθεί και οι αρχές ερευνούν τέτοια περιστατικά. Είναι αυτό μέρος της ε, πολιτικής κουλτούρας η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί εκεί πέρα από, με τρόπο φυσιολογικό και το να δημιουργούν προβλήματα στους δημοσιογράφους ή το οι δημοσιογράφοι να δορδοκούνται ήταν κάτι το οποίο ήταν στο παρελθόν αποδεκτό όσον αφορά τώρα τα ζητήματα των συνόρων υπάρχει ούτως ή άλλως ε, μια μεικτή επιτροπή που θα συνεδριάσει επίπεδο κρατών, ε, αρχηγών κρατών με την Κροατία και έχουν δηλώσει πως είναι διατεθειμένοι να προσφύγουν στη Χάγη. Και μετά υπάρχει το ζήτημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έχει χωριστεί σε Σερβική και Εκκλησία του Μαυροβουνίου. Αυτό προκαλεί ενόχληση στην κοινωνία, είναι υπαρκτό ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να λυθεί σε επίπεδο κράτους. Αυτό πρέπει να το βρουν οι εκκλησίες. Και να πω και κάτι άλλο είναι σημαντικό να μην ε, δημιουργηθεί ένα πεδίο παρέμβασης ε, στις σχέσεις ε, του άλλου κράτους. Μιλάω για Σερβία και Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο θα πρέπει να... Η Σερβία, με συγχωρείτε, θα πρέπει να σταματήσει να πιέζει τη το μοβούνιο μέσω της μειονότητας και των κομμάτων που περισσότερο προσανατολίζονται προς το Βελιγράδι. Ευχαριστώ. Κυρία Λούνα Τσακ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ για την έκθεση. Είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Εγώ θα αναφέρω τρία σημεία στα οποία θα ήθελα να Καταθέσει τροπολογίες και ελπίζω να τα στηρίξει ε, και ο συγητής. Για τα θετικά πρώτα απ' όλα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που λέει πρέπει το 2012 να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, το υποστηρίζουμε και αυτά για την ε, διαφθορά επίσης, αλλά υπάρχουν τρεις τομείς ε, στους οποίους θεωρώ πως θα έπρεπε να είναι πιο έντονη η έκθεση. Το ένα βεβαίως είναι περιβάλλον, ενέργεια, οικονομία, τα είπαμε και την τελευταία φορά για τον ποταμό στον οποίο σχεδιάζεται να γίνει ένα φράγμα. Ξέρετε πως ε, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες λίμνες των Βαλκανίων ε, που ε, έχει σημαντικό πλούτο βιοπικιλότητας. Εδώ πέρα λοιπόν θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό στη διαδικασία του διαγωνισμού να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να έχει μια στρατηγική για, τους, ε, για την υδροηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχω τίποτα κατά της υδροηλεκτρικής ενέργειας, αλλά θα πρέπει βεβαίως να σεβαστούμε και ε, τη βιοπικιλότητα που θα βοηθήσει και τον τουρισμό στη χώρα. Εδώ πέρα λοιπόν θα καταθέσουμε τροπολογία. Δεύτερον, κύριε Τάνοκ, ε, αναφέρατε κάποια πράγματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ε, αλλά δυστυχώς αφήσατε έξω τους ε, ΛΟΑΤ, λεσβίες, ομοφιλόφιλους κτλ. Και ξέρετε πως είναι αντιπροσωπεία και ο κύριος Κατσίν είχε πάει σε μια ημέρα κατά της ομοφοβίας, στην οποία έπεσαν δακρυγόνα και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα τι είχε γίνει. Η οργάνωση που την διοργάνωσε μάλιστα έπρεπε να δεχτεί η επίσκεψη της αστυνομίας στα γραφεία της. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη ε, ενημέρωση. Υπάρχει τώρα νόμος βεβαίως και ειδικό εντεταλμένος κατά των διακρίσεων αυτών, αλλά για την εφαρμογή αυτών χρειάζονται ακόμα κάποια βήματα και θα καταθέσω εδώ πέρα κάποιες τροπολογίες και το όσον αφορά τα δικαιώματα των φύλων μεταβατικών στην ε, νομοθεσία. Πρέπει να δούμε λοιπόν και την κατάσταση αυτής της ε, μειονότητας. Και εδώ πέρα καταθέσουμε τροπολογία. Και τέλος, μέσα μας και και ΜΜΕ ναι, υπάρχουν αυτά στην έκθεση, αλλά νομίζω θα έπρεπε να τονίσουμε περισσότερο τον ρόλο των ε, ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών, πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα δεν είναι δυνατόν ε, τμήματα της κυβέρνησης ή των αρχών γενικώ να κρύβονται. Και εδώ πέρα καταθέσουμε λοιπόν μια τροπολογία. Σε γενικέ γραμμέ, πάντω, συμφωνούμε με την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πως η υπόθεση της ενταξιακής διαδικασίας του Μαυροβουνίου είναι η πιο εύκολη περίπτωση από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Με αυτή την έννοια και η προσωπικά και μου που είναι υπέρ της ένταξης τελικά όλων των χωρών δεν έχει αντίρρηση η έκθεσή μας να προτρέπει για την έναρξη των ενταξιακών διαδικασιών. Όμως, σε σχέση με την έκθεση αλλά και την παρουσίαση του συναδέλφου, δεν ξέρω τι εννοούσε όταν είπε ότι χτες είδαμε διάφορους σουρεαλισμούς στη συζήτηση για το θέμα του κοσυφοπεδίου και για το θέμα της Φύρο. Αν σουρεαλισμό εννοούσε τα προβλήματα, τις εκκρεμότητες, τη σχέση με άλλες γειτονικές χώρες, τα προβλήματα του διεθνούς δικαίου. Εντάξει, στην περίπτωση του Μαυροβουνίου δεν έχουμε ευτυχώς τέτοια προβλήματα, η σχέση με τις γειτονικές χώρες, αλλά να μου επιτρέψει σε δύο σημεία παρακάτω ότι έχουμε άλλους σουρεαλισμούς ή τους λένε ρεαλισμούς της εποχής. Και θα σας πω ποιοι κατά τη γνώμη μου είναι αυτοί. Η έκθεση είναι εύκολη και κατά συνέπεια έχει την κλασική προσέγγιση μιας χώρας που θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτο σημείο. Από πότε η ένταξη ή η συμμετοχή ή το ΝΑΤΟ ως προθάλαμος θεωρείται κριτήριο για μια χώρα για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να τη δει κανείς ευνοϊκά. Αντιλαμβάνομαι τους ρεαλισμούς της εποχής, αλλά θέλω να σας πω ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι καθόλου δημοφιλές στην περιοχή, αλλά και είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν αποτελεί, όπως είπε χτες ο κύριος συνάδελφος, συγκολητική ουσία. Δεύτερο, το πρόβλημα τι ζητάμε σε μια χώρα όταν είναι στο προενταξιακό ε, καθεστώς, τι θα συζητηθεί στην περίπτωση που ανοίγουν οι φάκελοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, χτες στην Χτες στο Μαυροβούνιο, στην πρωτεύουσα, έγινε μεγάλη διαδήλωση. Με αιτήματα των διαδηλωτών κατά της λιτότητας. Τι χαιρετίζουμε σε αυτή την έκθεση. Χαιρετίζουμε το ότι ενσωματώνει τους κανόνες της ελεύθερης, όπως λέγεται, αγοράς. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης. Έχουμε δει τις αποτυχημένες συνταγές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς αυτούς τους κανόνες τους θεωρούμε ότι είναι ο μονόδρομος για την οικονομική πολιτική. Πού βρίσκεται η ανεργία λοιπόν, πού βρίσκονται το επίπεδο των μισθών, πού βρίσκεται το επίπεδο του κοινωνικού κράτους και το λέω αυτό όχι γιατί ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται σήμερα το Μαυροβούνιο, αλλά στις απαιτήσει, ας το πούμε έτσι τυπικά, στα οικονομικά κριτήρια της Κοπεχάγης όπως σήμερα ερμηνεύονται, πολύ φοβάμαι ότι προκειμένου να αποκτήσουν το ενταξιακό καθεστώς πάνε σε πιο σκληρά προγράμματα λιτότητας αδιαφορώντας για το επίπεδο της ανεργίας απλώς να πιαστούν κάποιοι δείκτες για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, οι μεγαλύτερες μας ενστάσεις, αγαπητοί συνάδελφοι και τελειώνω εδώ, είναι στο σημείο που αναφέρεται στο ποιες οικονομικές πολιτικές πρέπει να ακολουθηθούν, στην υποτίμηση των κοινωνικών προβλημάτων όπως ανεργίας και σε μια σειρά άλλα ζητήματα που ενδεχομένως συνδέονται και με αυτά, θυμίζω, νομίζω αυτό το αντιμετωπίζει, θα δω πιο ακριβώς την, πιο, με ακρίβεια την διατύπωση, διότι οι χτεσινοί διαδηλωτέ φώναζαν κατά μια διαφθαρμένης κυβέρνηση. Λοιπόν, Επομένω, το πρόβλημα της διαφθοράς θα το κοιτάξουμε πιο συστηματικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, άλλους Κούκαν, πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Μαυροβούνιο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους ε, προλαλήσαντες που έκριναν θετικά την πορεία του Μαυροβουνίου και να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ για την ε, έκθεση την ποιοτική που αξιολογεί αντικειμενικά και ρεαλιστικά την κατάσταση στη χώρα. Η χώρα προχωράει καλά στην πορεία της ένταξης και χαίρομαι για το ότι πέρσι έγινε ε, υποψηφίος ε, χώρα. Ελπίζω να συνεχιστεί η διαδικασία ομαλά και να ξεκινήσουν φέτος οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες και νομίζω σωστό είναι να ξεκινήσουμε με τα πιο δύσκολα κεφάλαια. Θα ήθελα έτσι να καλωσορίσω τον ορισμό του κυρίου Αλεξάνδρου Αντρέιπέιου ως διαπραγματευτή του Μαυροβουνίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις 7 προτεραιότητες ε, της έκθεσης του 2010 συμφωνώ με τον κύριο Τάνοκ πως είχαμε πρόοδο στο να τις ε, επιτύχουμε ειδικά στον αφορά το Κοινοβούλιο, το εκλογικό νόμο και τη χρηματοδότηση των κομμάτων, αλλά και σε βασικούς τομείς όπως η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης χαίρομαι για το ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον νόμο περί εκπαίδευσης των οποίων ε, πέρσι είχαμε μεγάλους πολιτικούς συμβιβασμούς. Όσον αφορά δε την ε, μείωση των ελλημάτων, ο προπολογισμός 2011 κινήθηκε εντός των κριτηρίων του Μάστριχτ. Το ότι εντάχθηκε στον ΠΟΕΔΕ το 2011 ήταν άλλη μία επιτυχία. Όλα αυτά νομίζω αποτελούν καλή αφετηρία για το Μαυροβούνιο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει και ελπίζω να κινηθεί προς σωστή κατεύθυνση. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα τομείς ε, που πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά. Πρέπει να, πρέπει να συνεχιστούν προσπάθειες στην καταπολέμηση διαφθοράς, ειδικά στα υψηλότερα επίπεδα και να παρακολουθούμε από κοντά τέτοιες περιπτώσεις όπως παραδείγματο χάρη ιδιωτικοποίηση τηλεπικοινωνιακών εταιριών. Επίσης συνεργασία του κράτους με την κοινωνία των πολιτών και εγγυήσεις για την ελευθερία των ΜΜΕ. Τέλος, ελπίζω το σχέδιο έκθεσης να αποτελέσει μια βάση για περαιτέρω συζήτηση και να βοηθήσει το Μαυροβούνιο στα επόμενα βήματά του στη διαδικασία ένταξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στους ε, υπόλοιπους συναδέλφους. Ε, παρακαλώ να παραμείνετε εντό του διλέπτου. Συνάδελφος Κάτσιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ για την πολύ καλά ε, ισορροπημένη έκθεση. Μιλώ εξ ονόματο ε, τη ε, πλειοψηφία τη Επιτροπή λέγοντα ότι προβλέπουμε στην έναξη των γεωργοτεύσεων με το Μαυροβούνιο τον Ιούνιο φέτο Το Μαυροβούνιο είναι μια μικρή χώρα και μια μικρή οικονομία αλλά από πλευρά ε, πολιτική αποτελεί παράδειγμα για τα υπόλοιπα Βαλκανικά κράτη για το πώ μπορούν να πετύχουν στη διαδικασία ένταξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ενθαρρυντικοί στο να ξεκινούν οι πραγματεύσει τον ε, Ιούνιο. Διότι όταν ξεκινούν οι πραγματεύσει με το Παραβούνιο, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στο Βαλκάνια όπω ε, όπως πριν. Το περιφερειακό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί γείτονε. Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Σερβία, Κωσυφοπέδιο, Αλβανία. Και αυτό θα είναι και ένα έναυσμα για την ε, Μακεδονία να ξεκινήσει διαπραγματεύσει και αυτή το συντομό των δυνατών. Ε, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και τη διαφθορά, Ε, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ελπισοπίας, θα πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις πτυχέ και να ε, φροντίσουν οι Μαροβούνοι να οδηγηθούν αυτές οι υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Οι διαπραγματεύσει ε, ένταξη είναι πολύ σημαντικέ σε ό,τι φορά την εφαρμογή του κράτου δικαίου. Όταν ξεκινούν οι διαπραγματεύσει, τότε θα είμαστε σε θέση να ε, προωθήσουμε τι ε, απαραίτητε μεταρρυθμίσει των δικαστικών κλάδων. Το βουνίο έχει κάνει καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση τη νομοθεσία τη σε πολλού τομεί. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω και κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό σχετικά με την ευρεία συνένεση στον τομέα της ε, εκπαίδευσης, της παιδείας και τα γλωσσικά ζητήματα. Ε, ε, χαίρομαι που υπάρχουν προσπάθειες για εξέβρεση συμβασμών προκειμένου να ε, καθησυχάσουν τις εντάσεις. Ελπίζω η έκθεση αυτή να μπορέσει να συμβάλλει με καλύτερη κατανόηση μεταξύ Βρυξελών, κράτα μέλη και της Ποργκόριτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συναλλούς Πέτερλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, κύριο Τάνοκ για την αντικειμενική αυτή έκθεση. Περιέγραψε τα πράγματα ως ε, έχουν, αλλά ξέρουμε πω το να είναι μικρή η χώρα δεν σημαίνει πω πρέπει να είναι και σύντομη η έκθεση. Η έκθεση είναι σύντομη γιατί το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει πρόοδο. Και αυτό σημαίνει πω έχει φτάσει η ώρα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Ελπίζω η χώρα να παραμείνει ε, τόσο δυναμική όσο είναι και να εφαρμόσει βεβαίως κατά του κράτους δικαίου και της οικονομίας αγοράς. Ο κύριος Τάνοκ για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ όλα τα σχόλια που άκουσαν ισχύουν την άποψή μου πως το Μαυροβούνιο είναι, σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ένταξή του και πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο Καλω ορίζω τα σχόλια του κυρίου Γκοαμφέρν πως πρέπει να κριθεί ε, από μόνο του βεβαίως αυτό τελώς και δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να υψώνουμε τον πύχη όσον αφορά την διεύρυνση. Ευχαριστώ και τη συναδελφή όσα είπαν και βεβαίως ε, αναμένω και την τις τροπολογίες των σοσιαλιστών και δημοκρατών για την κοινωνία των πολιτών, κατά πολέμηση της διαφθοράς κτλ. Όσον, αυτά, όσον αφορά αυτά τα οποία είπε ο κ. από τους φιλελεύθερους, τον ευχαριστώ και βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα οποία ξέρει και είπε για τις διαφορές των συνόρων ανέφερε και κάποιες συναντήσεις οποίες δεν ήξερα και ζητήματα μεταξύ της ε, Σερβικής ε, και ε, Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Εκκλησίας του Μαυροβουνίου. Νομίζω πως είναι κάπως ζητήματα πολύ λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να μας απασχολήσουν οι σχέσεις των δύο Ορθοδόξων Εκκλησιών. Κύριε Λούντσεκ, βεβαίω υποστηρίζω τη μεγαλύτερη διαφάνεια στους διαγωνισμούς, αλλά δεν θα υποστηρίξω τροπολογίες των πρασίνων που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας και το δικαίωμα τους ο κυρίαρχο να αποφασίσουν πώς θα έχουν ενέργεια. Αλλά βεβαίως δεκτές οι τροπολογίες σας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ. Όσον αφορά τον κύριο Χουντή από την ΚΟΕ, έκανε μια συγκεκριμένη αναφορά στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως ε, η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν είναι κριτήριο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι μια ένδειξη ε, όσον αφορά την οριμότητα και τη σταθερότητα της χώρας και δημοκρατικά και οικονομικά, ε, αν έχει και το ΝΑΤΟ εξετάσει την αίτησή τους. Δεν θα υποστηρίξω τη διαγραφή του ΝΑΤΟ από την παράγραφο Γ, νομίζω είναι στο εκτιμώντας Γ, γιατί αυτό απλά περιγράφει την εξωτερική πολιτική του Μαυροβουνίου και την στρατηγική τους. Δεν εξισώνω τον Άτομο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά αναφέρω πως ακολουθούν μια ευρωατλαντική κατεύθυνση στην εξωτερική της πολιτική και κύριε Βεβαίω πάντα καλωσορίζω αυτό το που έχει να πει. Είναι μεγάλος γνώμων στην περιοχή και στην εξωτερική πολιτική. Κύριε Κατσίν, βεβαίω δεκτά και τα σχόλιά σας. Και αν θέλετε να καταθέσετε κάποιες τροπολογίες ειδικά για τον ε, ρόλο του Μαυροβουνίου ως ε, μικρής χώρας, αλλά και όσον αφορά τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή στις διαφωνίες των γειτόνων του, ε, θα με ενδιαφέρει γιατί το έχω ακούσει αυτό στην Ποτγκόριτσα, πως θα ήθελαν ε, να ε, τοποθετηθούν ως ένας ουδέτερος διαμεσολαβητής μεταξύ άλλων χωρών στα Βαλκάνια και αυτό είναι κάτι το ενδιαφέρον και ο κύριος Πέτερ όπως και η κυρία Βρυσάγητς νομίζω σχολίασαν θετικά την έκθεσή μου. Ήμουν τυχερός που μου δόθηκε αυτή η έκθεση καθώς είναι κάτι το απλό νομίζω και εύκολο σχετικά. Αλλά βεβαίως αναμένω τις τροπολογίες σας και την τελική ψηφοφορία. Αλλά βεβαίως το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις των δυνατών. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω πως 2 ε, Φεβρουαρίου 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε στις 11 η ώρα. Με το σημαντικό ραντεβού που έχουμε προβλέψει οι αραβικές επαναστάσεις ένα χρόνο αργότερα και θα έχουμε προσκεκλημένους όπως τον ε, πρέσβευτή Τέιλορ και τον ε, πρέσβη Μπερναντήριο Λεόν αλλά και εθνικούς βουλευτές. Ευχαριστώ.

Συνάδελφοι, ώρα να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ενώπιόν μας ε, σχετικά με, τον, ε, με τις αραβικές επαναστάσεις ένα χρόνο αργότερα. Να καλωσορίσω τους συναδέλφους ε, και προσκεκλημένους έχουμε τους αξιότιμους φίλους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ επίσης να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να κάνουμε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση. Επαναλαμβάνω, το θέμα μας είναι οι αραβικές επαναστάσεις ένα χρόνο αργότερα. Νομίζω ότι είναι σημαντική η παρουσία των συναδέλφων από τα Εθνικά Κοινοβούλια, οι οποίοι συμμετείχαν και προτίθενται να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία που ενισχύει τις δημοκρατικές βάσεις της εξωτερικής μας πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, ε, με, σύμφωνα μάλλον με το πνεύμα της Εθνικής Λισαβόνας. Με αυτή τη συζήτηση το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να για μια ακόμα φορά την ε, σημασία που αποδίδει στις ε, σημαντικές αλλαγές ε, που τεκτενώνται στην ε, νότια όχθη της Μεσογείου. πριν από ένα χρόνο ο νησιακός λαός εξεγέρθηκε κατά του αυταρχικού καθεστώτος του Μπέναλη και ε, ανέλαβε την ευθύνη της, ανέλαβε την τύχη στα χέρια, τα χέρια του. Η διαδικασία της την προκάλεσε ε, μια πνοή η οποία παρέσυρε και άλλε αραβικές χώρες. Το εμβόλιο μας ήταν μεταξύ των πρώτων που εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτές τις εξελίξεις που μαρτυρούν ε, τη, μια νέα διάθεση των αραβικών λαών οι εξελίξει επέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάγκη μιας κατεπλήγουσα απάντηση και ανταπόκριση σύμφωνα με τις ιστορικές εξελίξεις και τα ιστορικά γεγονότα, αλλά τις υπόψη και τις ουσιαστικέ αλλαγέ που υπάρχουν μεταξύ των αραβικών αυτών κρατών. ήταν σημαντικό ω εκ τούτου για μα. να συζητήσουμε με τους ε, πολιτικούς πρωταγωνιστές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ξεκινήσουμε ένα κοινό προβληματισμό αναφορικά με τις άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις που οι αραβικές επαναστάσεις επιβάλλουν σε θέματα ασφάλειας, σταθερότητας και δημοκρατικής εξέλιξης των θεσμικών των οργάνων. Είναι σημαντικό είναι σημαντική και η αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκπροσωπείται σήμερα από τον πρόεδρο της Επιτροπής της Βενετίας, του οποίου η εμπειρία και οι νομικές ε, ε, μική πείρα που έχει θα μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο για τις εξελίξεις στην περιοχή. Να υπενθυμίσω ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας συμφωνούν με εμά ε, και επιθυμούν και αυτοί να δουν τις χώρες του Νότου του Μεσογείου να περάσουν αυτή τη φάση της ε, δημοκρατικής εξέλιξης και είναι μεταξύ μας ο πρέσβης William Taylor, τον οποίο και ευχαριστώ και η παρουσία του εντάσσεται στα το πλαίσιο συνεργασία που θα αποβεί προ όφελο όλων των εμπλεκομένων σε αυτή τη διαδικασία οικοδόμηση τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου στον αραβικό κόσμο. Οι λόγοι ανησυχία φυσικά δεν λείπουν και μια κοινή πολιτική προσέγγιση είναι απολύτω απαραίτητη. Κα, καταλήγω την ομιλία μου Ανοίγοντα τι εργασίε ε, για την πρώτη συζήτηση, της οποίας συντονιστή θα είναι ο συνάδελφο Πιέρα Αντώνιο Παντσέρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τους τρεις προσκεκλημένους μας τον κύριο Μπερναντίνο Λεόν, ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Νοτιού Μεσογείου, τον πρέσβη William Τέιλορ ειδικό συντονιστή για την ε, μετάβαση στην Εγγύς Ανατολή και τον κύριο Γιάννη Μπουμπίκιο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δημοκρατία, γνωστή ως Επιτροπή της Βενετίας. Αυτό το πρώτο τμήμα της ανταλλαγής απόψεων ε, νομίζω πως ε, θα μας δώσει την ευκαιρία να εξετάσουμε το ζήτημα από μια πραγματιστική πτυχή, με άμεση επαφή με την ε, πραγματικότητα της ε, μεταβατικής περίοδου. Υπενθυμίζω ότι και οι τρεις προσυκλημένοι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με εκπροσώπους ε, του Νοτιού Όχθης Μεσογείου σύμφωνα με την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ε, η εντολή του κ. Λεών εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων της νέας πολιτικής γειτονία προκειμένου να συνοδεύσουμε τους εταίρους μας του Νοτιού Τμήματος προς την δημοκρατική μετάβαση. Πολλές ε, πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει σε σχέση με τις χώρες εταίρους. Ε, θεωρίζομαι ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα τα οποία προέγυψαν μετά από τις πρώτες εκλογές και αναφέρουμε τις εκλογές στην Τινησία και την Αίγυπτο αλλά και τα όσα συμβαίνουν στην όλη περιοχή αλλά και τα πρόσφατα που φτάνουν από τη Λιβύη. Ναι. Η εντολή του πρέσβη Τέιλορ ε, ερμηνεύει και αυτό μια παρόμοια πολιτική βούληση που επιθυμεί να ακολουθήσει τις διαδικασίες ε, ε, και τις εξελίξεις στον ελληνικό κόσμο. Θέλει να μάθουμε περισσότερα για την αμερικανική στρατηγική σχετικά με την περιοχή και τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν αναλυφθεί τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ευχόμεθα φυσικά πως ο πρέσβης Τέιλορ να μας δώσει μια ανάγνωση των εξελίξεων που προέκυψαν στις αραβικές χώρες μετά από τις πρώτες εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Πολιτείες ε, ασχολούνται ο καθένας με τον τρόπο του και τη μέθοδό του και παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε πώς θα μπορούσαμε να συντονίσουμε τις ε, αμοιβαίες προσπάθειες και τέλος το Συμβούλιο της Ευρώπης συμμετείχε σε αυτήν την διαδικασία στήριξης της ε, δημοκρατικής ε, μετάβασης με την στήριξη της Επιτροπής της Βενετίας που είναι κάτι πολύ σημαντικό σε αυτή τη λεπτή φάση. Ο κ. Πουπίκιο που σας πενθυμίζω είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, της Βενετίας, βρίσκεται σε συνεχή διάλογο και επαφή με τους ε, πολιτικούς ε, ενδιαφερόμενους ε, και με τον ε, ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και με συνταγματολόγους. Η ανάλυση του λοιπόν, η ανάλυση των συνταγματικών και θεσμικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες όπως η Τινησία και η Αίγυπτος μετά από τις εκλογές, ε, τις νομοθετικές και τις συντακτικές στις δύο αυτές χώρες. Τελειώνω εδώ την ε, ομιλία μου. Θα δώσω το λόγο στον Περναντίνο Λεόν. Υπερθυμίζω στου ε, προσκεκλημένου ότι για να καταστήσουμε δυνατή μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχών στο σημαντικό σεμινάριο και είναι ε, δυνατότητα να υπάρξουν ερωταποκρίσει, θα ήθελα να δώσω 10 λεπτά σε έκαστο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σα ημέρα. Είναι Μεγάλη ευκαιρία για μένα το ότι βρίσκομαι ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα επιμείνει ευθύ εξ αρχή ε, πως ο διάλογος μαζί σα έχει μεγάλη σημασία και σκέφτομαι πως ε, μια που για τους νότιους μα. μας ε, ε, τα βασικά κέντρα εξουσίας είναι οι συντακτικές συνελεύσεις, τα νέα κοινοβούλια και επί τη ευκαιρία χαιρετίζω και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, νομίζω πως αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στον ρόλο μας ως εκπρόσωποι, στην επαφή μας με τις νέες αρχές. Η δική σας συστήριξη στήριξη, η συνεισφορά, ο διάλογος έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Νομίζω πως η συνεδρίαση, η σημερινή αφορά ιδιαίτερα το διεθνές πλαίσιο από τις ΥΠΑ, τους οργανισμούς, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο αυτό πολιτικό κοινωνικό πλαίσιο στην Νότια Μεσόγειο. Καμιά φορά αυτό βεβαίως αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά και αντιλαμβάνομαι πως αυτό ισχύει όταν ε, ε, διαβάζουμε διάφορες δημοσκοπήσεις, διαβάζουμε συχνά δημοσκοπήσεις ε, π.χ από την Αίγυπτο και γεγονό είναι πως όταν ρωτάνε τον κόσμο για διεθνείς εταίρους ε, η αλήθεια είναι πως η Ευρώπη δεν είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις ε, των ανθρώπων και υπάρχει αίσθηση πως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις χώρες πριν ε, αναλάβουμε δράση, πριν αποφασίσουμε για την μελλοντική μας στρατηγική και το μήνυμά μου είναι πως δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε εξαιρετικούς πόρους, η διεθνής κοινότητα έχει εξαιρετικούς πόρους στη διάθεσή της για να διαμορφώσει, να επηρεάσει το τι θα συμβεί στην περιοχή. Οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε θεατές. Πρέπει να έχουμε πλήρη συνεισφορά των ε, νομοθετικών ε, σωμάτων ε, και της εκτελεστικής εξουσίας και αυτό που πρέπει να κάνει και η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα. Με ρωτήσετε τώρα για πρωτοβουλίες διαλόγου με τις διάφορες χώρες μετά τις εκλογές, μετά τη διαδικασία στην κάθε χώρα να σχολιάσουμε το πώς βλέπουμε τις προκλήσεις στο προσεχές μέλλον και στο διεθνές πλαίσιο να αναφερθώ σύντομα στην κάθε χώρα της περιοχής. Πρώτα απ' όλα στην ε, την Ισία. Ξέρετε πως είχαμε μια ομάδα εργασίας και θέλω να το τονίσω αυτό όχι μόνο ε, με την κυβέρνηση της Ισίας αλλά με τα πολιτικά κόμματα, με την κοινωνία των πολιτών. Πολλοί εκπρόσωποι ε, είχαν εμπλακεί και έτσι μπορέσαμε να συνεργαστούμε και με τις νέες αρχές μετά τις εκλογές. Είχαμε λοιπόν τα τρία κόμματα, η Νάχτα, η ΠΙΑΡ και τα του σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ήταν στην ε, ομάδα αυτή εργασίας και βεβαίως προφανώς και μετά τις εκλογές ήμασταν σε στενή επαφή με τους επικεφαλείς αυτών των πολιτικών κομμάτων. Αύριο ταξιδεύω ξανά στην Τινησία. Θα δω τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τζαμπαλή. η δεύτερη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό αυτό μετά τις εκλογές. Η πρώτη η πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση ήταν μία-δύο ημέρες πριν του ζητηθεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, την οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε διάφορα ευαίσθητα ζητήματα και να δούμε την άποψή του για την συμφιλίωση το πώς θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με τους Ευρωπαίους Αμερικανούς, τη διεθνή κοινότητα και θα έχουμε νομίζω σημαντικά σημαντικές ειδήσει και μηνύματα από τον νέο Πρωθυπουργό της ε, Τινησίας και τις ιδιαίτερες σχέσεις που θέλει να έχει με την Ευρώπη. Μετά από την Τινησία θα γίνει άλλη μια συνάντηση της ομάδας εργασίας είναι πιο σημαντική ε, όσον αφορά την ενίσχυση των επαφών μας με τις νέες αρχές της Τινησίας όπου επιμένω ο ρόλος ε, του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι κρίσιμος Με την Ιορδανία, στην Ιορδανία έχω πάει ήδη πέντε φορές. Στις 11 ε, Φεβρουαρίου θα συναντηθώ με τον Βασιλιά, τον Αμπτουλάχ και πρέπει να πω πως ε, ήταν ε, πολύ εντυπωσιακή η συνεισφορά του όσον αφορά την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων κτλ. Και μπορώ να πω πως η Ορδανία από το Υπουργείο Εξωτερικών, ε, τον Υπουργό Σχεδιασμού κλπ. Ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θα ήθελα να τονίσω ε, δε τη συνεργασία μας ε, με τον Υπουργό Προεδρίας της ε, Κυβερνήσεως και τον αρμόδιο για την νομοθεσία που εμπλέκονται στη μεταρρύθμιση των επόμενων δύο-τριών μηνών που θα αποτελέσει νομίζω τη βάση για όλη αυτή τη διαδικασία. Στην δε τελευταία μας επίσκεψη συναντηθήκαμε με τα 11 κυριότερα πολιτικά κόμματα. Ήταν η δεύτερη φορά που υπήρχε η δυνατότητα να συναντήσουν την κυβέρνηση και προσεκλήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό τον ε, διάλογο. Στο τέλος δε της ε, συνάντησης εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων συμπεριλαμβανομένων πρέπει να πω και κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια συνάντηση που ήταν πολύ ειλικρινής, σκληρή μας είπαν οι εκπρόσωποι πως είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εκπρόσωπο διεθνούς οργανισμού σε αυτές τις άμεσες επαφές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την μετάβαση αυτή. Πέρα από αυτά τα 11 πολιτικά κόμματα είμαστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών όπως και στην Τινησία. Εγώ και η ομάδα μου συναντήσαμε πάνω από 20 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επόμενο βήμα είναι η ομάδα εργασίας μέχρι το τέλος ε, Φεβρουαρίου και νομίζω όπως και στην περίπτωση της Θηνησίας είχαμε σημαντική εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου ο Αντώνιο Παντσέρη και ο Ιγνάσιος Αλαφράνκα και ε, άλλοι ευρωβουλευτές ήταν παρόντες. Ελπίζω πως το ίδιο θα γίνει και στην περίπτωση της Ιορδανίας. Στην Αίγυπτο τώρα υπάρχει μια παύση, τελείωσαν οι βουλευτικές εκλογές, γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, θα ακολουθήσουν προεδρικές εκλογές ε, και μετά θα περάσει εξουσίες πολιτικούς. Ελπίζουμε οι Ισλαμιστές να συνασπιστούν με άλλες πολιτικές, ε, με άλλα πολιτικά κόμματα. Είμαστε σε στενή επαφή μαζί τους ε, Είμαστε λοιπόν σε επαφή με την ενδιάμεση κυβέρνηση, τις ε, αρχές, ε, οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών και πάλι εδώ πέρα με πολλές τέτοιες οργανώσεις. Στο Μαρόκο το ίδιο, προετοιμάζω το πρώτο μου ταξίδι μετά τις εκλογές. Έχω ήδη κάνει τρία ταξίδια εκεί και εκεί πέρα είμαστε σε πολύ στενή επαφή και θα ήθελα να τονίσω την σημασία των επαφών του Κοινοβουλίου μας με το Μαρόκο. Και είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα, να είμαστε σε επαφή. Ξέρω πως λαμβάνονται δύσκολες αποφάσεις σε σχέση με το Μαρόκο και επιμένω ε, επ' αυτού. Τέλος, για τη Λιβύη θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, 30 και 31 Ιανουαρίου. Ένα, μια συνάντηση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΟΗΕ, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Δούνο του ε, έχουμε την ευθύνη για τον συντονισμό όλων των προσπαθειών της διεθνούς ναι. κοινότητας και όλες οι χώρες οι εμπλεκόμενες ε, θα εκπροσωπηθούν ε, από τους τρεις αυτούς οργανισμούς και αναμένω να οργανώσουμε και μια συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών ε, κατά πάσα πιθανότητα τον Φεβρουάριο για να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με τη Λιβύη, να προετοιμάζουμε τις εκλογές που είναι βεβαίως ο βασικός στόχος αλλά και για να μπορέσει να επανέλθει η ομαλότητα σε τομείς κρίσιμους, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλεια διαχείριση συνόρων κλπ. Σύντομα τώρα, για τις προκλήσεις όπως ανέφερα και σε προηγούμενες παρεμβάσεις, ε, τα οικονομικά και τα πολιτικά πρέπει να κινούνται από κοινού. Οι διαδηλώσεις αυτές αφορούν βεβαίως την αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια έχει μια πολιτική διάσταση. ελευθερία, βεβαίως δικαίωμα, οι εκλογές, αλλά και οι δουλειές, οι θέσεις εργασίας ε, είναι πάρα πολύ κρίσιμες και βεβαίως απαιτείται από την ε, διεθνή κοινότητα να φροντίσει οι χώρες αυτές να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν κάτι και να έχουν οικονομίες που λειτουργούν. Οπότε να τονίσω πως το μίσο, πως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η γεωργία είναι μίσο κλειδιά εάν θέλουμε οι οικονομίες αυτές να λειτουργήσουν. τις πολιτικές πτυχές νομίζω πως ε, ο διάλογος, ε, περισσότερος διάλογος είναι σημαντικός με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να οικοδομήσουμε ε, γέφυρες. Αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο θεσμικά αλλά και κοινωνία ως κοινωνία στο επίπεδο το ανθρώπινο και εγώ επιμένω πως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Οι χώρες αυτές αλλάζουν δραματικά, αλλά και εμείς πρέπει να αλλάξουμε, να αντιληφθούμε διαφορετικά το τι συμβαίνει. Πρέπει τεχνικά να εμπλακούμε σε όλες τις μικροδιαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, ε, οι νομοθετικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούν ε, ισχυρή παρουσία και βεβαίως όσον αφορά την παρατήρηση των εκλογών. Να σας πενθυμίσω εδώ πέρα την έκθεση Γκάλερ για την Τινησία που έγινε δεκτή με τρόπο θετικό. Επίσης για τον πρέσβη τον κύριο Τέιλορ που βρίσκεται εδώ πέρα σήμερα παρόν είναι ικανός διπλωμάτης ε, και Βεβαίω, συνεργαζόμαστε και με τη ΣΥΠΑ και με τον ΟΗΕ και με διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και με χώρες του κόλπου, με την Τουρκία ε, και την Ελβετία, Κίνα, Νότια Κορέα, Νορβηγία, ακόμα και το Ισραήλ που θέλουν να εμπλακούν στις διαδικασίες αυτές και να συνεργαστούν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές της Νοτιού Μεσογείου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο πρέσβης William Taylor. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η παρουσία μου εδώ μπροστά σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για την παρουσία του φίλου μου Βερναρδίνου Λεόν. την ευθύνη αυτή την, και το ενδιαφέρον μας για τις μεταβάσεις αυτές στις χώρες εκείνες τις παίρνουμε πολύ σοβαρά. Πρέπει να βρούμε πόρους, βρήκαμε και χρειάζεται κάποια οργάνωση αυτών των μεταβάσεων, των μεταβατικών διαδικασιών. Όπως είπε και ο Βερναρδίνο, πρέπει να στηρίξουμε και τη Λιβύη και την Τινησία και την Αίγυπτο και ο Βερναρδίνο πρόσθεσε δύο χώρες, το Μαρόκο και την Ιορδανία, που εγώ δεν έχω ως ευθύνη. Οι μεταβάσεις αυτές, οι μεταβατικές διαδικασίες στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθούν και ελπίζω στο σύντομο μέλλον, εκτός από τις τρεις χώρες, την Ισία, Λιβύη και Αίγυπτο, θα προσθεθούν η Εμένη και η Συρία στον αριθμό των χωρών που κινούνται προς τη δημοκρατία. Πιστεύουμε, συμμεριζόμαστε δηλαδή την πεποίθηση ότι πρόκειται για το σημαντικότερο γεωπολιτικό συμβάν από το 89 και θέλουμε να στηρίξουμε τις διαδικασίες αυτές όσο μπορούμε. Εμείς στα Συνωμένα Πολιτείας θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν τη στήριξη των μεταβατικών διαδικασιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια επιρροή εκεί και γι' αυτό πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών οι εμπορικές η πολιτική γειτονίας, οι σχέσεις που έχετε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές και η ηγεσία που επιδείξατε στην καμπάνια του ΝΑΤΟ για τη Λιβύη δείχνουν πόσο σημαντική θα ήταν για μας η συνεργασία με σας. Πήραμε μαθήματα για τη σταθερότητα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η πραγματική σταθερότητα, η βιώσιμη σταθερότητα, η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή αυτή δεν θα προέλθει από την υποστήριξη ε, αυταρχικών καθεστώτων. Κάναμε στο παρελθόν λάθη και αναγνωρίζουμε ότι η πραγματική σταθερότητα προέρχεται από κυβερνήσεις που κυβερνούν με τη συνένεση του λαού τους σημαντική έννοια αυτή που την παίρνουμε πολύ σοβαρά όπως και εσείς. Και θέλουμε αυτήν την έννοια να στηρίξουμε τώρα στην περιοχή εκείνη. Συνένεση των διοικουμένων σημαίνει και δίκαιες και αδιάβλητες εκλογές και οργάνωση θεσμών που να είναι υπόλογοι προς τους πολίτες. Είναι σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων μειονοτήτων γυναικών που είναι σημαντικά συστατικά στοιχεία αυτού της, της ενίας. Θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα της δικαιοσύνης και της ενόμου τάξεως ή του κράτους δικαίου. Θεωρούμε ότι αυτές είναι ανθρώπινες αξίες που τις ζητούν οι Άραβες όπως και οι Ευρωπαίοι, όπως και οι Αμερικανοί, είναι κοινέ αξίες. Κοινέ μεν αξίες, αλλά σε, διαφορετικό, σε διαφορετικά συμφραζόμενα και πλαίσια. Στην Τινησία φαίνεται ότι που ήταν ο ηγέτης και χρονολογικά αλλά και πολιτικά των εξελίξεων αυτών, γιατί εκεί άρχισε η ε, Αραβική Άνοιξη, εκεί έγιναν οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές, που όλοι τις θεώρησαν δίκαιες και αδιάβλητες, και ο συνασπισμός που προήλθε από αυτές συμπεριλαμβάνει και το κόμμα Εναχντά που θεωρείται Ισλαμιστικό, σε συνεργασία με κοσμικά κόμματα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Τινησίας προτίθενται να κάνουν την πρώτη τους διεθνή επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι. Δείχνει ότι αναγνωρίζουν, σέβονται και εκτιμούν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναζήτησή τους της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Υποστηρίζουμε πλήρως και τις οικονομικές και τις πολιτικές εξελίξεις όπως είπε και ο Βερναρδίνος γιατί αυτά τα δύο συνδέονται δεν μπορεί το ένα να πετύχει χωρίς το άλλο ενώ αν πετύχουν και τα δύο μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Προτείναμε λοιπόν και επεξεργαζόμαστε εγγυημένα δάνεια ενθαρρύνουμε τον ιδιωτικό τομέα και αμερικανικές επιχειρήσεις και αναδυόμενες επιχειρήσεις στην Τινησία και ένα από τα κυριότερα διεθνή προγράμματα που εφαρμόζουμε είναι το λεγόμενο Peace Corps το οποίο λειτουργούσε και στην Τινησία την εποχή του Μπεναλή και συνεχίζει τώρα η από την Ισιακή καθοδήγηση. Στην Αίγυπτο τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δυναμική εκεί και πάλι υπήρξαν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και πάλι το Ισλαμιστικό κόμμα Ελευθερία και Δικαιοσύνη κέρδισε και ένα άλλο κόμμα και αυτό Ισλαμιστικό οι σαλαφιστές δηλαδή, επίσης τα πήγαν πολύ καλά. Και αναμένουμε ότι το τινησιακό πρότυπο θα εφαρμοστεί και στην Αίγυπτο. Θα δούμε τι θα κάνει ο συνασπισμός και πώς θα καταφέρουν να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί. Αναγνωρίζουμε πάντως πάλι και εδώ τη σημασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και τις ανθρώπινες αξίες. η δέσμευση του στρατού να παραδώσει την εξουσία σε πολιτική κυβέρνηση είναι επίσης πολύ θετική εξέλιξη. Η αλλαγή του συντάγματος που το συνέγραψε μια επιτροπή εκατομελής επίσης είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία την οποία υποστηρίζουμε Καλύτερα βέβαια να οι εξελίξεις να είναι ταχύτερες. Θα δούμε τι θα κάνει λοιπόν η καινούργια κυβέρνηση. Η κοινωνία των πολιτών της Αιγύπτου επίσης εξελίσσεται γοργά. Την υποστηρίζαμε και στο παρελθόν και συνεχίζουμε να την υποστηρίζουμε και τώρα και οικονομικά και επικοινωνιακά και μέσω των πολιτικών κομμάτων. Όπως και οι Ευρωπαίοι, έχουμε πολιτικές οργανώσεις που δεν υποστηρίζουν μεμονωμένα κόμματα, αλλά την ανάπτυξη της πολιτικής ζωής γενικότερα. Δυστυχώς, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση πολλές από αυτές τις οργανώσεις που υποστήριζαν γενικότερα την ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων και όχι μεμονωμένα κόμματα, ε, επιτέθηκε εναντίον τους και κατά Αιγυπτιακών και Ευρωπαϊκών μήκη όμικρων. Αυτό είναι πρόβλημα και για τους Αιγυπτίους και για μας, γιατί εμείς θέλουμε αυτές οι μήκη όμικρον να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν και οι υπολογιστές τους και τα άλλα περιουσιακά τους στοιχεία που κατασχέθηκαν να επιστραφούν για να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν ελεύθερα. Και όσο το περιμένουμε αυτό θα υπάρχουν δυσκολίες όσο δεν έχει λυθεί. Παρ' όλα αυτά υποστηρίζουμε την Αίγυπτο δηλαδή δίνουμε σημαντική στρατιωτική βοήθεια που είναι ιδιαίτερα εκτιμάται ιδιαίτερα από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση και για πρώτη φορά φέτος ε, αυτό αναφέρθηκε επίσημα καθώς και η όροι της. Τώρα η Λιβύη. Εδώ υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και δυσκολίες για την, για την οργάνωση των εκλογών, πράγμα το οποίο και αυτό υποστηρίζουμε. Στην Τινησία και στην Αίγυπτο ξέρουμε λίγο πολύ πώς οργανώθηκαν οι εκλογές Στη Λιβύη όμως δεν ισχύει αυτό, είναι μεγάλη πρόκληση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι στηρίζει τη διοργάνωση των εκλογών αυτών, των εκλογικών διαδικασιών. Επίσης υποστηρίζουμε όπως είπα και πριν την Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία και ηγεσία στο θέμα της στήριξης της Λιβύης Χαιρόμαστε που ο ρόλος μας είναι απλώς βοηθητικός όπως κάναμε και στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Θα συντονιστούμε με τον ΟΙΕ για να συνδυαστεί και η δική μας και η δική σας βοήθεια. Και τέλος, γενικότερα περιφερειακά, χαιρόμαστε που μπορούμε να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που άρχισαν πέρυσι οι Γάλλοι θα συνεχίσουμε δηλαδή την εταιρική σχέση της Ντοβίλ. Η Προεδρία μας τον Μάιο θα συνέλθει στο Σικάγο για να προωθηθούν να συνεχιστούν αυτά που ταυτίστηκαν τότε στην Ντοβίλ ως προς τη συνεργασία με επενδυτές, επενδύτριες και την κοινωνία των πολιτών. Αναμένω τώρα τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι πρόκειται για την ευκαιρία του αιώνα Ευρωπαίοι και Αμερικανοί να συνεργαστούν για να πετύχει η Αραβική Άνοιξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Και τώρα θα ακούσουμε την άποψη της ε, Επιτροπής της Βενετίας μέσω του Πρόεδρου του κυρίου Τζάνι Μποτικιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βρέθηκα στην Τινησία προέτους, το Μάρτιο, με τον ε, τέος πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο και ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξο, όπως εξάλλου και ο ίδιος ο πρόεδρος μετέβην και την περασμένη εβδομάδα, αλλά η αισιοδοξία μου δεν ήταν η αυτή δεν είναι ότι είμαι λιγότερο αισιόδοξο ε, για την Τινησία, αλλά και για τι υπόλοιπε Αραβικέ χώρες. Αλλά από την άλλη πλευρά λέω ότι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χρειάστηκε πάνω από 20 χρόνια για να ολοκληρώσει την ε, δημοκρατική μετάβαση και δεν ε, κατάφεραν όλοι να φτάσουν σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Τώρα, ε, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να πανεμποδιστεί ε, όλε τι διαδικασίε δημοκρατικέ. Πρώτα απ' όλα για την Τινησία το ζήτημα είναι οικονομικό. Εάν δεν βοηθήσουμε την Τινησία σε οικονομικό επίπεδο με, το εκατο, με τα εκατομμύρια των ε, ανέργων ε, που θα έχουμε φέτος, ένας αριθμός ο οποίο αυξήθηκε σημαντικό μετά από την πόλεμο στη Λιβύη, που οδήγησε 150.000 ε, στην Τινησία, άνεργους ε, και λόγω του ότι πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λόγω της αστάθειας ε, της πολιτικής ε, έλλειψη ασφάλειας κοινωνικών διεκδικήσεων κλπ. αποσύρθηκαν από την, την, την αγορά. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει λοιπόν είναι μια κοινωνική έκρηξη για οικονομικούς λόγους. Κατά τα υπόλοιπα τα πράγματα πάνε καλά. Για το Μαρόκο δεν είναι τόσο το οικονομικό ή κοινωνικό πρόβλημα που προέκυψε, αλλά οι καθυστερήσεις, οι χρονοτριβές σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της, ε, του, του συντάγματος ε, και λένε ότι το Δημοκρατικό Σύνταγμα στο Μαρόκο θα χρειαστεί τουλάχιστον μία θητεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διάστημα αυτό. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις για την εφαρμογή του συντάγματος στο Μαρόκο να γίνουν το των δυνατών. Τώρα για την Αίγυπτο υπάρχουν μια σειρά προβλήματα, υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα, η Αίγυπτος είναι σημαντική χώρα και πληθυσμιακά αλλά και για το πολιτικό βάρος που έχει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά μετά από τις πρόσφατες εκλογές είχαμε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι προς όφελος της δημοκρατίας, οι αδελφοί μουσουλμάνοι και οι σαλαφίστες που πήραν 17% ε, ενώ οι αδελφοί μουσουλμάνοι το 44% θα έχουν λοιπόν την συντριπτική πλειοψηφία στην Βουλή και αυτή η πλειοψηφία θα είναι πολύ ισχυρή με τους, την παρουσία των δύο αυτών κομμάτων. Αυτή είναι η άποψή μου για την Αίγυπτο. Για τον Μπαχρέιν ε, παραδείγματο χάρη χώρα για την οποία δεν μιλήσαμε, αλλά μόνο τα αυτά γνώρισε κινήματα σημαντικά, ετίθεται το θρησκευτικό ζήτημα. Η περίσχυση των Σιητών επί της ε, πλειοψηφία των Σουνιτών είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει και στη Συρία κατά την άποψή μου και θεωρώ ότι πολλές αραβικές χώρες ε, ε, κοιτάνε τα τεκτονόμενα στην Συρία και ειδικά την πτώση του καθεστώτος των Χαλαβητών, αλλά κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ρήξη για τον άξονα των συζητών στην περιοχή. Ξεκινάει από τη Συρία και καταλήγει στο Μπαχρέιν. Αυτά λοιπόν όλα με κάνουν να είμαι πιο απεσιόδοξο από την προενός έτους, αλλά λέω παράλληλα ότι θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο. Η δημοκρατία δεν οικοδομείται μέσα σε μερικούς μήνες ή σε λίγα χρόνια. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σας είπα ότι χρειάστηκαν πολύ περισσότερους χρόνο. Πιστεύω ότι οι αραβικές χώρες έχουν μια ευκαιρία διότι υπάρχει ένα πολιτιστικό επίπεδο ανώτερο από το που υπήρχε στις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ε, με την κατάρρευση του στίχους. Υπάρχει μια ιτελιγέντσια που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την δική μας. Υπάρχει μια κοινότητα των πολιτών που είναι ισχυρή σε πολλές από αυτές τις χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά θα διευκολύνουν την ε, ενίσχυση της δημοκρατίας και την παγιωσή της. Επανέρχομαι τώρα στην Τινησία και στο νομικό πλαίσιο, διότι ξέχασα να σας πω πως η Επιτροπή της Βενετίας, για όσους δεν τη γνωρίζουν, είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος, συμβουλευτικός του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δρά στον επίπεδο του συνταγματικού δικαίου. Μετά από την κατάρρευση του τύπου του Βερολίνου, ε, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βοηθούμε όσες δημοκρατίες το επιθυμούν να αναθεωρήσουν τις δημο... τα συντάγματά τους και να τα εναρμονίσουν με τα οικουμενικά πρότυπα της δημοκρατίας. Η Επιτροπή της Βενετίας ε, τα είχε ιδιαίτερη διορατικότητα διότι ακούσαμε, ε, συναισθηθήκαμε το, το κλίμα και επιθυμίας ε, αλλαγής ε, από το 2006 στις αραβικές χώρες. Το 2006 αρχίσαμε τις επαφές αρχικά με την ε, Αλγερία, το Μαρόκο, την Τινησία, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν και τη Λιβύη. Και όλα αυτά ενώ τις επαφές δεν έγιναν με τις, επαφές, με τις αρχές, αλλά στο Συμβούλιο το Αραβικό μέσο, θα έλεγα, του νομοθετικού συστήματος ε, που υπήρχε στα κράτη αυτά, μεταξύ των οποίων ε, ε, προσώπων υπήρχαν άνδρες και γυναίκες που επιθυμούσαν περισσότερη δημοκρατία. Από το 2006 λοιπόν ξεκίνησαμε τις επαφές μας. Πολλοί από τους έγιναν πλήρη μέλη της Επιτροπής Βενετίας όπως το Μαρόκο, Αλγερία, την Ισία, Αίγυπτος ήθελε να γίνει μέλλον, το επιθυμεί ακόμα, αλλά λόγω της καταστάσεως που επικρατεί στη χώρα θα χρειαστεί κάποιο χρόνος. Η Παλαιστινική Αρχή έχει ένα ειδικό καθεστώς, έχουμε πει και το Ισραήλ. Υπάρχει, είναι λοιπόν ένα φόρουμ, επιτροπή μας, ε, στο οποίο έχουμε συγκροτήσει και μια υποεπιτροπή για την νότιο όχθη της Μεσογείου. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει στι αρχές Μαρτίου και θα συζητήσουμε με τους Άραβες συναδέλφους μας ε, θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Δεν την ουσία λοιπόν το νομικό πλαίσιο είναι σταθερό και εξελίσσεται προς το στην κατεύθυνση. Τελικά μπόρεσαν να κάνουν αυτό που επιθυμούσαν. Οι εκλογές ε, μετατέθησαν για μερικούς μήνες και αυτή η συντακτική συνέλευση ε, συγκροτήθηκε, ξεκίνησε τι εργασίε της. Ε, απέκτησε ένα είδος ε, μικρού συντάγματος και στόχος είναι να ε, συντάξει ένα σύνταγμα εντός ενός έτους, αλλά δήλωσαν ευθύς εξ αρχής ότι επειδή έχουν την ε, λαϊκή νομιμότητα, η συμφωνία που είχε επιτευχθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της Επιτροπής Σούερ που είχε δημιουργήσει τις βάσεις για την συγκρότηση αυτής της συντακτικής συνέλευσης δεν ισχύουν άρα θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο και θα εργαστούν ε, κατά το δοκούν. Αλλά όλες οι επαφές ε, που είχα στην Τινησία, όλα τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν φυσικά στην ε, συντακτική συνέλευση, με διασφάλισαν πως δεν θα τους χρειαστεί πάνω από 18 μήνες και οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν τον Άνοιξη του 2013. Το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν προχωράει, υπήρξε ε, πρόβλημα για την υιοθέτηση του στρούγγανισμού του συνέλευσης, αλλά επιλύθηκε το πρόβλημα την πέσμενη εβδομάδα. Την, ε, υπήρχε ένα πρόβλημα για τη σύνθεση των 7 επιτροπών που θα σαλαμοποιήσουν ε, το διαδικασία κατάρτιση συντάγματος και θα δουλέψουν για ένα ενίο πρόγραμμα ε, υπάρχουν 7 επιτροπές, είναι μια συντονιστική που παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο και την οποία ο Μπεν ο πρόεδρος της συντακτικής συνέλευσης, ήθελε να λάβει την προεδρία. Ε, από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν έχω περισσότερε πληροφορίε. Ε, υπήρθε κάποιο συμβασμό. Ο Μπεν Τζαφάρ θα λάβει την Προεδρία και οι 7 επιτροπέ θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους άμεσα. Λοιπόν, από νομοθετικής πλευρά τα πράγματα προχωρούν. Η εκλογική επιτροπή, η οποία είχε συγκροτηθεί για αυτές τις εκλογές, λειτουργήσε σωστά, εκτός από την συγκρότηση των εκλογικών καταλόγων, διότι 57 μόνο ή 52% του εκλογικού σώματος ε, καταχωρήθηκε που δεν είναι στο κόμμα του Ναντά θεωρούν ότι το Νάντα δεν έχει το 34% των εκλογικού σώματο, αλλά μόνο το 18% διότι 34% του 52%. Ε, σε επόμενε εκλογέ λοιπόν, αν όλοι εγγραφούν στου εκλογικού καταλόγου και αν όλοι ψηφίσουν, τότε το Ναντά που ε, πήρε του περισσότερου ψήφου, γιατί είναι και το πιο πειθαρχικό ψαχημένο κόμμα θα υποχωρήσει και θα αφήσει χώρο στους υπόλοιπους. Διότι η Τρόικα, δηλαδή τα τρία κόμματα που συμμετέχουν στον συνασπισμό στο πλαίσιο της συντακτικής συνέλευσης έχουν μια άνετη πλειοψηφία που δεν είναι των δύο τρίτων αλλά είναι ε, παραπάνω από την απόλυτη πλειοψηφία που είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση αυτής της νομοθεσίας αυτού του οργανικού νόμου. Και το Σύνταγμα θα πρέπει στο σύνολο να εγκριθεί από τα δύο τρίτα, αλλά ε, το, η τελική ψηφοφορία για, για τα άρθρα θα πρέπει να έχει 7 ψήφους παραπάνω. Τώρα αυτά ε, ο, κύλησε ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου. Θα στο Μπαχρέιν να πω ότι υπάρχουν κάποιες ε, κινήματα, κάποιες κινήσεις ε, για μια διεθνή συνεργασία και για να προσπαθήσουν να αλλάξουν τη χώρα, όπως και στην Ιορδανία, όπου γίνονται ε, επαφές μεταξύ Συμβούλου της Ευρώπης και της Ιορδανίας για μια επικείμενη επίσκεψη για την συγκρότηση ενός κοινού πρόγραμματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση, να περάσουμε στις, ε, στη συζήτηση. Κλείνουμε εδώ τον κατάλογο των παρεμβάσεων. 15 συνάλφοι μου ζητήσει το λόγο. Έχουμε φυσικά και ζητήματα από τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και από το Ευρωκοινοβούλιο. Για λόγους, ε, θα έλεγα, αυρότητας θα ήταν καλύτερο να κάνουμε μια θετική διάκριση, αν συμφωνείτε, για τους ε, συναδέλφους που ρώνονται από τα κράτη-μέλη και θα τους ε, δώσουμε δύο λεπτά για κάθε παρέμβαση. έως εκ τούτου, 1,5 λεπτό θα χρειαστεί να μιλήσει κάθε ένας εξήμων των Ευρωβουλευτών. Εν αλλάξει λοιπόν ε, θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Κυρία Ανταλάρα έχει το λόγο από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, και θέλω εδώ να εξάρω την πρωτοβουλία σας για ακόμη μια φορά να καλέσετε τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτή την τόσο κρίσιμη συζήτηση ε, και ανταλλαγή απόψεων και να πω εδώ ότι συμφωνώ απόλυτα με την παρέμβαση του κυρίου Λεόν. Ε, I endorse, Mr. Leon, the coherent relation και δέχομαι και εγώ κύριε Λεόν την αναγκαιότητα που υπάρχει μιας, ενός συντονισμού μεταξύ Ένωσης Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών. Μια στάθεια. Τα όσα συνέβηκαν τελευταία δεν είχαν προβλεφθεί από τη διεθνή κοινότητα παρά το γεγονός ότι πολλοί σημείωναν την ανάγκη διασφάλισης αρχών δημοκρατίας και διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Βέβαια, καμία περίπτωση δεν είναι η ίδια με την άλλη. Είδαμε χθε τα γεγονότα πάλι στη Λιβύη Υπάρχει όμως μια κοινή συνισταμένη η απέτηση των λαών της περιοχής για περισσότερη δημοκρατία και ίσες ευκαιρίες στην πρόοδο και στην ανάπτυξη, αλλά και ένας εσωτερικός ανταγωνισμός συμφερόντων των μεγάλων παικτών στην περιοχή. Γι' αυτό στο λίγο χρόνο που έχω θα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι εποχή και είναι πολύ νωρίς να ζητήσουμε την κεφαλαιοποίηση αυτών που παρενέβησαν στα αραβικά κράτη. Είναι πολύ νωρίς κύριοι συνάδελφοι. Στις έκτακτες συνθήκες η διεθνή κοινότητα καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διαχειριστεί αυτή τη διεθνή κρίση που έχει δυνητικά ε, επικίνδυνες προεκτάσεις για το χυμαζόμενο Νότο και για την πατρίδα μου την Ελλάδα. Γι' αυτό όποιες πρωτοβουλίες παρθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην αποφυγή της διόγκωσης των φαινομένων μετανάστευσης, την αποφυγή της δημιουργίας αιστιών έντασης που θα ανακυκλώνουν τη βία, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, την παροχή υλική και τεχνικής βοήθειας, ώστε οι χώρες αυτές να μπουν σε, τροχιά σταθερότητας. Τέλος, τη διασφάλιση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών που έχουν σχέση με τα κράτη-μέλη στις χώρες αυτές. Ειδικότερα, η κατάσταση στη Συρία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η βία φέρνει περισσότερη βία. Πρέπει να κινηθούμε με προσοχή γιατί οι περιφερειακές συνέπειες στην περίπτωση της Συρίας μπορεί να είναι εξαιρετικά αποσταθεροποιητικές για το σύνολο της Μέσης Ανατολής. Ένα όμως είναι σαφές. Το καθεστώς Ασάντ με την πολιτική καταστολής και ομής βίας που ακολουθεί παίρνει ένα δρόμο χωρίς γυρισμό. Γι' αυτό οφείλει να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα. Μετά, η διαιώνιση του Παλαιστινιακού επηρεάζει τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή. Οι Παλαιστίνοι πρέπει να αποκτήσουν επιτέλους την πατρίδα που δικαιούνται. Οι Ισραηλινοί πρέπει να ζήσουν επιτέλους τις συνθήκες ασφάλειας που επίσης δικαιούνται. Η λύση θα προέλθει από ειρηνευτική διαδικασία. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η Ευρωπαϊκή Διπλωματία πρέπει να διασφαλίσει ότι αντί μια σύγκρουση πρέπει επιτέλους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι εφικτό. Δεν είναι μόνο η κρίση η οικονομική που απασχολεί τα μέσα. Η Ελλάδα έχει παραδοκισιακές σχέσεις φιλίας με την Παλαιστίνη και μια νέα ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με το, Ισραήλ, αλλά και στενές σχέσεις με όλες τις χώρες. Με όχημα αυτό πρέπει να πορευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω ότι αν μακρηγορείτε αυτό οδηγεί στο να περιορίσετε ή και να απαγορεύσετε σε κάποιους συνάδελφο να λάβει το λόγο. Και αυτό δεν είναι πολύ ευγενικό. Κυρία Άννα Γκόμες, 1,5 λεπτό να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Eh, eh, e Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τους δύο ομιλητές. Ελπίζω ο κύριος Λεόν να εντυπωσιάσει και να επηρεάσει και την κυρία Άστον για την επόμενη σύνοδο. Γιατί όσο υπάρχει εσωτερική κρίση στην Ευρώπη δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αποτελεσματικοί εκτός αυτής. Η σταθερότητα είναι απαραίτητη και στις δύο περιοχές, την Αραβική και την Ευρωπαϊκή και άλλη, υπάρχει αλληλεξάρτηση. Θέλω να ρωτήσω όμως τον πρεσβευτή Τέιλορ. Στην Τινησία τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ένωση οικονομικά για να βοηθήσει τη χώρα. Στη ΔΕ τι γίνεται εκεί ως προς την οργάνωση της πολιτικής ζωής. Ίσως γίνουν εκλογές, δεν ξέρουμε όμως πώς οργανώνονται πολιτικά τα κόμματα. Υποστηρίζουμε επαρκώς την κοινωνία των πολιτών, τις γυναίκες, βοηθούμε τους Λίβιους να δημιουργήσουν έναν σωστό δικαστικό τομέα. Ε, Και επίσης για τον πρεσβευτή Τέιλορ. Τι μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε για να πιέσουν το στρατό στην Αίγυπτο ώστε να συμβαδίζει με τις δημοκρατικές αρχές η λειτουργία του. Ξέρω ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της Αιγύπτου γενικότερα και για την ειρνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν το αγνοώ. Και η χώρα που δεν αναφέραμε είναι η Αλγερία. Τι φρονείτε για την Αλγερία και το Μαρόκο και ο ΕΜΕΝ και ο ΔΕ. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφο Γκέιπ, ε, Βουλή των Εκπροσώπων. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο Αμερικανός μας συνάδελφος. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στον αραβικό κόσμο πρέπει να νοηθεί ως ολόκληρη διαδικασία, όχι σαν ένα μεμονωμένο γεγονός και θα χρειαστούν μάλλον δεκαετίες ολόκληρες πριν μπορέσει να λειτουργήσει μια πραγματική πλουραλιστική κοινωνία στις χώρες αυτές. Μερικές χώρες θα προχωρήσουν περισσότερο, άλλες λιγότερο. Και ξέρουμε και από ευρωπαϊκές χώρες που παρατηρούμε και αυτή τη στιγμή ακόμα ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στον εκδημοκρατισμό και στη δημιουργία ενός μια συνταγματικής τάξης και του δικαστικού τομέα. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν τι λέμε. Ταυτόχρονα πρέπει να θέσουμε μερικά ερωτήματα και προβλήματα ιδιαίτερα στην, ε, στο μανιφέστο 93 σελίδων της μουσουλμανικής αδελφότητας γιατί περιέχει μερικά στοιχεία που θα αποτελέσουν τεράστια προβλήματα και θα ήθελα να σχολιάσετε την εξωτερική πολιτική της Αιγύπτου και τι θα μπορούσε να γίνει, ποιο θα ήταν το μέλλον της ε, συνθήκης της με το Ισραήλ μετά τις εκλογές. Τώρα επειδή δεν έχω πολύ χρόνο θα ήθελα να περιοριστώ στο ότι πρέπει να προσέχουμε επίσης πώς χορηγούμε τη βοήθεια στις χώρες της Βόρειας Αφρικής φαίνεται ότι δίνουμε χρήματα χωρίς όρους με μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας και σε δικτατορίες με τρομερές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ τώρα βάζουμε όρους στις χώρες που κινούνται προς τη δημοκρατία. Αυτό θα μπορούσε κανείς όντως να το πει ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά αλλά πρέπει να βάλουμε βέβαια όρους αν θέλουμε να εφαρμοστούν οι πανανθρώπινες αξίες για τις οποίες μίλησε ο πρεσβευτής Τέιλορ. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πώς τα βλέπουμε όλα αυτά και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο θα το προσέξουν πάρα πολύ να μην υπάρξει ξένη παρέμβαση. Ευχαριστώ ε, κύριο Μιλανμόν για 1,5 λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεόν για τα λόγια του. Νομίζω ότι αυτή η είδηση που μας έδωσε είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική. Θα πρέπει εμείς να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις όπως το πράττουμε από πέρυσι τον Ιανουάριο. Τότε είχαμε επικρίνει κάποιες καθυστερήσεις ε, της κυρίας Άστον. Βλέπω ότι ο κύριος Λεόν έχει αρχίσει να τα τροποποιεί όλα αυτά, να αλλάζει τα ασφάλματα του παρελθόντος. Θα πρέπει λοιπόν να ομολογήσουμε ότι αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα όπως ε, αυτό των πολιτικών κομμάτων ε, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες έχουμε και ελάχιστες σχέσεις και επαφές. Τώρα, Τώρα ε, βλέπουμε ότι στο Αιγυπτιακή Βουλή την πλειοσοφία την έχουν οι ε, Ισλαμικά κόμματα. Ε, πριν από τρεις μήνες υπήρχε μια, υπήρξε μια task force ε, που ασχολήθηκε με το ζήτημα των ε, κοινωνικών εξελίξεων και ε, συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Γκόμες για την Αλγερία. Είναι μια χώρα που βρίσκεται πολύ πλησίων, έχει σημαντικούς ενεργειακούς πόρους, είναι πολύ σημαντική θέση της και δεν αναφέρθηκαν οι τρεις προσκεκλημένοι μας καθόλου σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Νίρεστάιν. Τέλος. Η Συνάδελφο, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω και από τους τρεις αγορητές το εξή. Έχω την εντύπωση ότι εδώ αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον όρο σταθερότητα. Αλλά νομίζω ότι είναι σφάλμα να επαναλάβουμε ένα λάθος του παρελθόντος. Καταρχήν ε, δώσαμε τη δυνατότητα μια σταθεροποίηση στην Ασία και την Αφρική με σχέσεις ε, με τους δικτάτορες. Τώρα δεν θα ήθελα να, απο... να φροντίσουμε μόνο την βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και όχι τις δημοκρατικές εκλογές. Κάτι το οποίο πολλές φορές οδηγεί σε περαιτέρω αστάθεια Οποιοδήποτε γνωρίζει την ε, ιστορία του Ισλάμ ξέρει ότι το ιδεολογικό κομμάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο πλευρά μα θα ήταν θεμελιώδε λάθο να κρίνουμε ότι να αγνοήσουμε αυτέ τι ε, συνθήκε ε, σημαίνει ότι τους πρόκειται προς την αντίθετη κατεύθυνση της δημοκρατίας. θα ήθελα λοιπόν να με διαφωτίσετε και κάτι ακόμα. Ήδη από πλευρά μα ο όρο ε, Αραβική Άνοιξη αντικαταστάθηκε από όρου πιο γενικού, ε, εξέγερση, επανάσταση, ε, κάτι το οποίο μα προβληματίζει. Φυσικά έχουμε, θα, εκφράζουμε το θαυμασμό μας για όσους διαδήλωσαν στις πλατείες και στους δρόμους κατά των δικτατόρων που επί δεκαετίες καταπίεζαν τους λαούς αυτούς. Ε, ε, φυσικά εγώ δεν θα ήθελα να αναφέρω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Αυτό το οποίο κάνουμε με επισκέψεις, συναντήσεις, ε, συμφωνίες, συνθήκες κλπ. είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε το δρόμο της δημοκρατίας. Άρα είναι δύσκολο να εντοπίσουμε με ποιο τρόπο μπορεί να ακολουθεί αυτή η οδός της δημοκρατίας. διαπιστώνουμε ότι ενώ στο παρελθόν με κάποιες ομάδες που είχαν ε, απογορευτεί από τα τότε καθεστώτα ε, απέκτησαν ε, την υποστήριξη των λαών των καταπιεσμένων και σήμερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αυτές οι ομάδες λοιπόν φέρουν ένα όνομα αυτό του εξτρεμισμού των Σουνιτών είτε πρόκειται για αδελφότητα είτε φέρουν κάποια άλλα ονόματα. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να αντικαταστήσουμε τον ε, πανεραβισμό από τον ε, ε, Ισλαμική αδελφότητα. Θα πρέπει λοιπόν να μην αφήσουμε να γίνουν αυτές τις εξελίξεις. Αν ξέρετε την ιστορία της Ισλαμικής αδελφότητας γνωρίζει πολύ καλά και ολοκληρώνω πρόεδρε. Θα κάνουμε συμφωνίες. Θεωρώ λοιπόν πως η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει υποστήριζοντα τα δικαιώματα των γυναικών, τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα ε, και να μην διεξαχθεί πόλεμος με το Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να σας πω. Πασχολήσω. Ευχαριστώ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, και εγώ όπως ε, και πολλοί άλλοι από του παρεμβαίνοντε ε, έχω απογοητευτεί από την πορεία που έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμή η Αραβική Άνοιξη, ειδικά στην ε, Αίγυπτο και βεβαίω δεν χύνουμε δάκρυα για την πτώση των τυράννων, αλλά παρόλα αυτά η εκλογή του Αλνούρ στην Αίγυπτο είναι ιδιαίτερα ανισχυτική και φαίνεται πω η Άνοιξη γίνεται αραβικό χειμώνα και αντί για να έχουμε κάτι ανάλογο με το τείχος του Βερολίνου. Φοβάμαι πως ζούμε κάτι ανάλογο με το 1979, την πτώση δηλαδή του Σάχη του Ιράν, την οποία ακολούθησε για λίγο ένας μετροπαθής ηγιώτης και μετά ένα μεσαιωνικό θρησκευτικό καθεστώς που είναι τώρα αποφασισμένο να αποκτήσει πυρνικά όπλα. Και τώρα πρέπει να πω πως το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο που έχει 67% και παραπάνω Ισλαμιστές με ανησυχεί και το ερώτημά μου προς τον πρέσβη τον κύριο Τέιλορ είναι θα προτείνατε να σταματήσουμε άμεσα κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την ε, Αίγυπτο εάν απομακρυνθεί από την ε, στρατηγική του Camp David και την ειρήνη με το Ισραήλ. Επίση στην Συρία κανεί βεβαίω δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον κοσμικό με ένα αλλά δικτάτορα δεν Μπασάρ Αλασάντ. Αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται πάλι καθορίζουν την πορεία οι Ισλαμιστές οι οποίοι ε, θα επιβάλλουν φοβερά αντίπεινα στους ε, χριστιανούς εάν ε, λάβουν ποτέ την εξουσία. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Και βέβαια το άλλο ερώτημα για εμένα είναι το μήπως θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε την εξωτερική μας πολιτική υπό το φω. Ε, του ότι ακραία κόμματα καταλαμβάνουν την εξουσία σε χώρες κλειδιά όπως η Αίγυπτο και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις μετριοπαθείς μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες παρά το ότι δεν είναι δημοκρατίες παραμένουν πυλώνες σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή. Ευχαριστώ, συνάδελφος Κλίχ από την Πολωνική Βουλή. Ε, χάθηκα, χάρηκα ιδιαίτερα για αυτά τα οποία είπε σήμερα και ο κύριο Σουλεόν και ο πρέσβης ο κύριος Στάιλερ γιατί μας δείχνει πόσο διαφοροποιημένη προσέγγιση μπορούμε να έχουμε ε, για το πώς μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς οι προσεγγίσεις των ΙΠΑ και της Ευρώπης, αλλά είναι ευέλικτες και μας δίνουν περισσότερες επιλογές γιατί ε, η Αραβική Άνοιξη δεν ήταν κάτι το ενιαίο ή ένα ομοιογενές ε, γεγονός το πώς εξελίχθηκε. Οπωσδήποτε στην Αίγυπτο και την Τινησία είχαμε μαζικά κινήματα, αλλά στη Λιβύη παραδείγματο χάρη ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Ο Καντάφη δεν έφευγε χωρίς ε, δεν θα έφευγε χωρίς ε, την στήριξη του ΝΑΤΟ παραδείγματο χάρη. Και νομίζω πως ε, στη Συρία παρόμοια θα είναι η κατάσταση. Χωρίς στρατιωτική εμπλοκή δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Κατόπιν οι Ισλαμικές δυνάμεις και τα κινήματα τα οποία αναφέραμε. Ο κύριος Τάνοκ σωστά λέει πως ο στρατός για χρόνια κρατούσε σε απόσταση τα ριζοσπαστικά Ισλαμικά κινήματα και νομίζω πως ε, δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά δημοκρατικά αφελείς και να μας συναρπάζουν οι δημοκρατικές διαδικασίες γιατί η δημοκρατία χωρίς κάποιες φιλελεύθερες απόψεις, η δημοκρατία η οποία βασίζεται μόνο στην διαδικασία δηλαδή μπορεί να οδηγήσει στην γέννηση πιο ε, ακραίων ε, ισλαμιστικών κινημάτων. Όσον αφορά τη λεγόμενη ε, οικοδόμηση θεσμών, ε, ακούμε πάρα πολλά πράγματα, ακούμε διαφορές για το πώς θα πρέπει εμείς να εξάγουμε δημοκρατικές αξίες. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό νομίζω είναι να ξανασκεφτούμε την οικονομική μας εμπλοκή στην διαδικασία ανοικοδόμησης σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα αφού υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες σε αυτή την περιοχή, γιατί αν δεν στηρίξουμε την δημοκρατία θα ξαναγυρίσουμε στα παλιά και ισλαμιστικά. Σας ευχαριστώ, κύριος Πέτερλε. <clears throat> Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους τρεις ομιλητές για τις αφίστους τους παρουσιάσεις. Αν ήθελα να μιλήσω σαν γιατρός που κάνει διάγνωση θα έλεγα ότι η πρώτη αυτή φάση τελείωσε της ακρόασης δηλαδή. Υπήρξαν μεγάλες προσδοκίες αλλά και πολλή απογοήτευση. Όλες αυτές οι κοινωνίες δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μόνες τους τον δημοκρατικό τους δρόμο και συμφωνώ με τον κύριο Λεόν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο πρέπει να σκεφτούμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας και να αρχίσουμε αμέσως διάλογο με κοινή εξέβρεση λύσης και με πνεύμα εταιρικής συνεργασίας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές και ότι αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε πώς θα σεβαστούμε τις διαφορές αυτές. Δέστε τι γίνεται με τις διώξεις χριστιανών και στην Ιγυρία, όχι μόνο σε αυτές τις χώρες. Πρέπει λοιπόν να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας προοδευτικά, όχι με μιας όπως κάνουμε συνήθως. Πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε την κοινοβουλευτική διάσταση της συνεργασίας, να βρούμε δηλαδή νέες μεθόδους για να τονίσουμε ποια θεωρούμε ότι είναι τα βασικά προβλήματα της περιοχής. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε για την Κύπρο. Thank you. Uh, I share the concerns expressed uh, the Arabs not to be turned out. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις ανησυχίες για το πώς uh, μπορεί η Αραβική Άνοιξη να καταλήξει Αραβικός χειμώνας. Μόνο από την διαδικασία για δίκες και αδιάβολητες εκλογές. Τα θέματα ασφάλειας θα πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα μας. Ήδη στις δύο χώρες που έγιναν με δίκες και αδιάβολητες εκλογές, οι Ισλαμιστές εξασφάλισαν την πλειοψηφία. Και χθε παρατηρήσαμε την εκλογή μέλους της Ισλαμικής Αδελφότητος ως πρόεδρο του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, οι δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες να μην καταλήξουν εξελιχτικά σε καθιστώτα τύπου Ιράν. Είδαμε τι έχει συμβεί στο Ιράν μετά την ανατροπή του Σάχη. Και ένα δεύτερο και τελευταίο μου σχόλιο. Δημοκρατία χωρίς οικονομική, δημοκρατία χωρίς οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία δεν μπορεί να υπάρξει. Την ίδια ώρα η δημοκρατία από μόνη της δεν μπορεί να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Molto bene, grazie. Σας ευχαριστώ. Ο συνέρφος Αρλάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν η Αραβική Άνοιξη, το εάν θα, η Άνοιξη θα γίνει αεροϊκός χειμώνας εξαρτάται και από εμάς. Εμείς ε, υποστηρίζαμε όλα τα προηγούμενα καθεστώτα και αν θέλουμε να επηρεάσουμε τη διαδικασία πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στην πραγματικότητα. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υποστηρίζουμε τα δημοκρατικά καθεστώτα ε, τα υποστηρίζαμε όταν ε, κατερεάν, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε αρκετά θετικοί για διάφορα βασίλεια, εμμυράτα, ε, τα οποία έχουν πάρα πολύ καταπιεστικούς μηχανισμούς και εξακολουθούμε να τους πουλάμε και όπλα. Αναφέρομαι ειδικά στις ΙΠΑ, κύριε Πρέσβη. Λέτε πως κάνουμε λάθη στο παρελθόν, αλλά τώρα ακολουθούμε το σωστό δρόμο κτλ. Αλλά εξακολουθείτε να πουλάτε πάρα πολλά όπλα στα φεουδαρχικά αυτά καθεστώτα, Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, Μπαχρέιν. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική είναι περιοχές όπου ανθεί ε, το εμπόριο όπλων και τους δίνουμε τα μέσα για να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτον. Και δεύτερον, Εγώ θα έλεγα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ δεν ε, έχουν ακόμα αξιόπιστες συνεκτικές πολιτικές σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ. Ε, Madame Arena, κυρία Αρένα από την Βελγική Γερουσία. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Pour l'occasion qui nous euh, Μας δίνεται σήμερα μια ευκαιρία να παρεύουμε πάνω στα ζητήματα αυτά. Να πω ότι η πολιτική γειτονία που χρησιμοποιήθηκε χθε δεν είχε όρου και προποθέσει. Πάντω, εγώ χθε είδα ότι υπήρχαν προποθέσει οικονομικέ σε ό,τι την πρόταση σε πόρου, προποθέσει μεταναστευτικού χαρακτήρα, και να δούμε τι συμφωνίε που είχαν υπογραφεί με τη Λιβύη για να. Ε, για τα θέματα τα μεταναστευτικά ή ακόμα και κάποιες προϋποθέσεις ε, αντι-Ισλάμ. Θα πρέπει λοιπόν να μην επαναλάβουμε τέτοιου είδους προϋποθέσεις. Άκουσα διάφορα πράγματα για τη μετανάστευση, ε, ίσως ε, άλλη μία ε, προϋπόθεση αντι-Ισλάμ. Θα πρέπει λοιπόν ως Ευρωπαίοι να δουλέψουμε πάνω σε νέες προϋποθέσεις, νέους όρους και να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Θα πρέπει λοιπόν, να προτείνω όρους που άπτονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, την εγγύηση όλων των δημοκρατικών εξουσιών, δηλαδή μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αλλά να ευνοήσουμε και τη συνεργασία νότου-νότου. Η Ευρώπη δούλεψε πολύ σε επίπεδο διμερών σχέσεων με κάποια κράτη, ε, συνεργασία η οποία όμως απέβαινε εις βάρος ε, της ε, συνεργασίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με χώρες του Νότου, δηλαδή Νότους-Νότους. Και ως γυναίκα θα ήθελα να ζητήσω να υποστηριχθούν όλες οι κοινωνίες των πολιτών και ιδιαίτερα οι γυναικείες. Ευχαριστώ. Επόμενος, επόμενη ώρα, η κυρία Βίλαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία. Πρώτον, έγινε μία ενδιαφέρουσα σύγκριση της περιοχής αυτής με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω έναν τομέα ιδιαίτερα όπου η Ευρώπη καθυστέρησε πολύ στην στήριξη δηλαδή πολιτικών κομμάτων και της οικοδόμησης αυτών. Αν συγκρίνουμε με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα θυμηθείτε όλοι πόση υποστήριξη είχε δοθεί στα καινούρια αναδυόμενα πολιτικά κόμματα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Τουλάχιστον οι φιλελεύθεροι έχουν στείλει παρατηρητές εκεί στις χώρες, στις αραβικές χώρες από το Σεπτέμβριο και πρέπει αυτό να το πάρουμε πιο σοβαρά υπόψη μας. Και το δεύτερο μου σχόλιο είναι ερώτημα δηλαδή και προς τους δύο μιλητές, τους πρεσβευτάς Λεόν και Τέιλορ. Αφορά τη συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία στην περιοχή και την βοήθεια που εκείνη χορηγεί τι σχόλια έχετε να κάνετε γι' αυτό. Πώς σχολιάζετε δηλαδή τη συνεργασία των χωρών αυτών ιδιαίτερα της Συρίας αλλά και άλλων με τη Ρωσία. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Κρόφοντ από τη Δανία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική εισαγωγή. Είπα ήδη πως ε, πρέπει να αφήσουμε πίσω την ε, παλιά πολιτική, ότι δηλαδή υποστηρίζαμε την σταθερότητα και όχι την αλλαγή. Θεωρούσαμε πως ε, μια σταθερή δικτατορία ήταν καλύτερη από απρόβλεπτη αλλαγή. Τώρα πλέον έχουμε νέα δεδομένα και ανάλογα πρέπει να κινηθούμε. Οπότε δεν ε, νομίζω πως πρέπει να μας προξενεί έκπληξη το ότι στην Τινησία και στην Αίγυπτο κέρδισαν οι Ισλαμιστές. Ήταν ε, αυτοί στο παρελθόν στην αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε στήριξη στην κοινωνία των πολιτών ε, πολύ πιο ενεργά. Είναι μέρος της νέας μας πολιτικής γειτονίας, το ανέφερε ο κύριος Λεόν. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν περισσότερα πράγματα στον τομέα αυτών. Τα πιο κοσμικά κόμματα, μη θρησκευτικά, ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν έχουν και στήριξη. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τη, την οικοδόμηση νέων κομμάτων, των συνδικάτων και άλλων ομάδων. Είναι μεγάλη μεταβατική περίοδος και δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει το ότι οι εκλογές, ε, οι, οι πρώτες εκλογές ε, ε, πήγαν στους Ισλαμιστές. θα μπορούσαμε επίση να δούμε τον τομέα τη ε, οικονομία και μέσω τη ανάπτυξη ο κόσμο να στρέψει τα νότα του στου Ισλαμιστές. Οπότε το ζήτημα είναι πώ θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη στήριξή μα για την κοινωνία των πολιτών και θα ήθελα να ακούσω την άποψή για τι συνταγματικέ διαδικασίε που έχουμε στην Αίγυπτο και αλλού. πώ θα μπορέσουμε mm. εκεί να διασφαλίσουμε ε, διαδικασίες οι οποίες θα σέβονται τα οικουμενικά δικαιώματα. Σας ευχαριστώ κυρία Φλότρα. Ε, ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τους ομιλήσαντες και τονίζω ιδιαίτερα αυτά που είπε ο πρεσβευτής Τέιλορ, δηλαδή ότι κάναμε λάθη, είπε. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι οι δικτατορίες εγγυώνται σταθερότητα και ο... καταλάβαμε ότι η ανάπτυξη είναι αναπόσπαστη με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοινοτοπίες βέβαια ακούγονται όλα αυτά, αλλά είναι βασικά. Γιατί πράγματι οι κοινωνίες των πολιτών δεν καταλαβαίνουν ποια ακριβώς είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον λέει ότι ανέκαθεν εμείς υποστηρίζαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ πρόκειται δηλαδή για δοκιμή στα μάτια τους της δυνατότητάς μας να πάρουμε στα σοβαρά υπόψη αυτές τις αλλαγές στις αραβικές χώρες. Υπάρχει το θέμα της συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι εκεί υπάρχει μεγάλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τίθεται το ερώτημα ακόμη κι αν υπάρχει τυπικά στήριξη στις πολιτικές διαδικασίες, τι γίνεται εάν το καθεστώς είναι θεμελιωδώς διεφθαρμένο. Υπάρχει και το θέμα της μετανάστευσης, αλλά η κινητικότητα και το δικαίωμα του πηγαινοέρχεσθε είναι και αυτά βασικά. Δεν χρειάζεται πια θεώρηση για να πηγαίνει κανείς στην Τινησία, αλλά για να έρθουν οι Τινήσοι τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα. Δεν πρέπει υψοφάκτο να θεωρούμε ότι συστηματικά η μουσουλμανική αδελφότητα στην Αίγυπτο θα κάνει θα συνεργαστεί με τους σαλαφιστάς και σαλαφίστριας ο κυβερνών συνασπισμός δεν έχει συνάψει σταθερές συμμαχίες μέχρι τώρα και το έχει αποδείξει σε πολλές του ψηφοφορίες ότι μπορεί να δεχτεί να χάσει εξουσία παρά να κάνει ορισμένες συμμαχίες. Δεν είναι δεδομένα όλα αυτά δηλαδή. μπορεί να κάνουν και άλλου είδους συμμαχίες από αυτές που αναμένουμε. Κύριε Τέιλορ, μιλήσατε για τη Συρία, αλλά αν μπορείτε να μας πείτε τίποτε παραπάνω, θα σας ήμασταν ευγνώμονες. Κύριος Γκάλε. Επικεφαλής της αποστολής μας στην Ισία. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το ότι δεν Σα άκουσα από την αρχή. Αναφερθήκατε στην αποστολή μου και σα ευχαριστώ. Όσον αφορά την Τινησία τώρα, όπως είπε και η κυρία Φλότρ, νομίζω πως έχουμε μία πιθανότητα ω Ένωση δεδομένου του μεγέθου τη χώρα και του πλαισίου που είναι σχετικά θετικό, έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε κάποια πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με ενθαρρύνει, παραδείγματο χάρη, όταν κάθεσα και την έκθεσή μου στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τζαμπαλή, στις 6 Ιανουαρίου, καλώς όρισε την παρουσία μας ε, αφενός με την αποστολή τεχνικής αρρωγής που βρίσκεται επί τόπου και μπορεί να βοηθήσει την συντακτική συνέλευση στο έργο της και την κυβέρνηση σε κάποια ζητήματα, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την ε, θετική τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα και στον οικονομικό τομέα, συγκεκριμένα στην ε, την Ισία. Γιατί αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι σε έναν μηχανισμό, ενός, ε, σε ένα συνασπισμό ενός μετριοπαθούς Ισλαμικού κόμματος με τα κοσμικά κόμματα να έχουν αποτελέσματα γιατί αυτό θέλει ο κόσμος δεν έχει πλέον υπομονή και για να αποφύγουμε αυτή την αυτοεκπληρούμενη ε, προφητεία από οι ακραίοι θα καταλάβουν την εξουσία, ειδικά στην Τινησία πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο γρήγοροι και συγκεκριμένοι για να βοηθήσουμε τη νέα αυτή κυβέρνηση για να εμπιστευτούν τη νέα δημοκρατική κατάσταση οι άνθρωποι και εκεί πέρα νομίζω έχουμε πιθανότητες να επιτύχουμε. 30 δευτερόλεπτα στον συντονιστή κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ. Μεταξύ των όσων ακούσαμε υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία στην όλη μας συζήτηση σχετικά με το ρόλο και τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δερματίσουν ε, τις εξελίξεις Εμεί εδώ εκπροσωπούμε διάφορα θεσμικά όργανα, αλλά αποτελούμε και την έκφραση πολιτικών κομμάτων. Πιστεύω ότι η δυνατότητα στις ε, χώρες που εμπλέκονται στην Αραβική Άνοιξη ε, ότι θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερο πλουραλισμό είναι αν συμβεί με την ε, εξέλιξη και ανάπτυξη των λαϊκών κομμάτων. το θέσμα της πολιτικής συνεργασίας είναι αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, κάτι το οποίο συνοδεύει την πολιτική γειτονία. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του Δ. Μπουκίκιο πάνω στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα για τις απαντήσεις, καθένας από εσά οι θα έχει 6 λεπτά στη διάθεσή του. Πολύ σύντομα στην κυρία Νταλάρα, κάθε άστο μίλησε για τα τρία μη. Για... Ε, με στόχο δε μεταξύ άλλων την κινητικότητα. Η μετανάστευση λοιπόν αποτελεί σημαντικό μέρος στρατηγικής μας. Αναπτύσσουμε στρατηγικές κινητικότητας με το Μαρόκο, την Αίγυπτο, την Τινησία και με τους Ιορδανούς. Ε, αυτό. Ε, προς την κυρία Αναγκόμες. Βεβαίω συμφωνώ πως η ασφαλειά τους είναι και η ασφαλειά μας και δεν εργαζόμαστε μόνο διμερώς αλλά και μέσω μιας περιφερειακής προσέγγισης Ντοβίλ, G8, Ένωση, Μεσογειακή. Ε, δεν ε, ασχολούμαστε λοιπόν μόνο με αυτές τις μικροδιαδικασίες αλλά σε μια ευρύτερη προοπτική και συμφωνώ πλήρως. Τι κάνουμε τώρα στη Λιβύη. Αυτή η συνάντηση που έχουμε τώρα, 30 και 31 Ιανουαρίου, θα ασχοληθεί με ζητήματα κλειδιά για να ξεκινήσει μια ομαλοποίηση στον οικονομικό, στον πολιτικό, στον κοινωνικό τομέα. Συνεργαζόμαστε στενά με την κοινωνία των πολιτών και τις ερχόμενες εβδομάδες θα αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που αναφέρατε και τα πολιτικά κόμματα, ενώσεις γυναικών, πολιτικές ενώσεις, παρατηρήσεις εκλογών και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τον κύριο, προς τον κύριο Γκέιτς. Θα συνεργαστούμε με τις νέες αυτές ε, πολιτικές δυνάμεις επί τη βάση αρχών και μεταξύ αυτών των αρχών βεβαίως είναι πολλά ζητήματα σημαντικά για τις διεθνείς σχέσεις, η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πολύ υψηλά σε αυτές τις προτεραιότητες. Επισκέφθηκα το Σεπτέμβριο το Ισραήλ, ανταλλάξαμε απόψεις ε, για τη στρατηγική που έχουμε στην περιοχή και επιμένω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Τώρα για την αιρεσιμότητα, του διαφορούς όρους, συμφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει να φροντίσουμε πως κανείς δεν θα πιστοχωρήσει. Ε, δεν ε, αμφισβητεί κανείς ε, βεβαίως την δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το τι συμβαίνει και να φροντίσουμε πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο μέλλον. Για τον κύριο Μιγιάν, ε, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, η κυρία Άστον και όλοι εμείς ε, βεβαίως εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά. Όχι μόνο από την σκοπιά της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αλλά λαμβάνοντας πάντα υπόψη ε, και αυτά τα οποία λέει το Κοινοβούλιο, ο κύριος Μπρόκο, ο κύριος Σαλαφράγκα είναι αναμειγμένοι στην ε, υπόθεση αυτή. Τώρα όσον αφορά την Τουρκία είναι σημαντικό να εμπλακεί ε, είναι σημαντική οικονομία με ανάπτυξη και είναι υπόδειγμα για αυτές τις χώρες. Βεβαίως, όλες, όλοι θέλουμε οι χώρες αυτές να είναι επιτυχείς και άρα το τουρκικό μοντέλο θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίω πολλές από αυτές οι χώρες είναι κοντά στην Ευρώπη με πολλούς τρόπους και Ήδη πολλοί πρωθυπουργοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να έρθουν κοντά στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα την Τινησία, πράγματι έχετε δίκιο, υπάρχει ανησυχία για, τις εξεγέρσεις κτλ. Η Αλγερία είναι σημαντική χώρα και κάνει βήματα, θα έλεγα, προς σωστή κατεύθυνση. Προσπαθεί να βρει τη θέση της στη διεθνή σκηνή, να βελτιώσει τη σχέσεις της με το Μαρόκο, να ανοίξει περισσότερο πολιτικά μιλώντας, αλλά δεν είναι ε, μία από τις χώρες ε, που βρίσκεται σε μετάβαση. Αλλιώς, ε, εντάξει, οι σχέσεις μας με την Αλγερία, εμπόριο κτλ. είναι φυσιολογικές, αλλά πρέπει να σημειωθεί πρόοδος, αλλά δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή άμεσα με την Αλγερία. Όσον αφορά τώρα τις αρχές ε, και τα δικαιώματα, νομίζω πως εδώ πέρα, εάν δείτε τα Ισλαμικά κόμματα, πρέπει να θυμάστε πως όλα έχουν και εθνικιστικό πρόγραμμα, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και Υπάρχει βέβαια και αυτά τα οποία είπε ο κ. Τάνοκ ε, για τη Συρία. Η Συρία όμως δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή μέρος της εντολής μας. Εμείς ασχολούμαστε με τις υπόλοιπες χώρες που επηρεάστηκαν από την Αραβική Άνοιξη. Ε, δεν υπάρχει τίποτα τώρα που να μπορώ να πω αυτή τη στιγμή για το καθεστώς της ε, Συρίας όσον αφορά τις ε, χώρες ε, του κόλπου. Πρέπει να διατηρήσουμε την υφιστάμενη εξωτερική πολιτική. Δεν βλέπω λοιπόν, να αλλάζει εκεί πέρα η πολιτική. Ε, κάπου πάμε. Καλά, κάπου αλλού όχι τόσο, έτσι για να απαντήσω όπως τον κύριο Κλής, αλλά θα πρέπει νομίζω να παραμείνουμε συνεπείς με τους ε, στόχους μας για τα σχόλια του κυρίου Πέτελε. Τώρα συμφωνώ πράγματι πως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία μια περιφερειακή προσέγγιση. Έχουμε την Ένωση της Μεσογείου, τις 18 αυτές χώρες ε, και πρέπει να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για κάθε ομάδα χωρών είπε κάποιος από εσάς πως ε, δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία χωρίς ανάπτυξη. Πράγματι προσπαθούμε να ενθερύνουμε την ανάπτυξη και κατόπιν την ε, δημοκρατία και κατόπιν προς τον κύριο Αρλάκη. Κοιτάξτε, για να είμαστε αξιόπιστοι έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας, αλλά έχω την εντύπωση πως όλες οι χώρες που είναι σε μετάβαση νομίζω πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση και για τα σχόλια της ε, κυρίας Αρένα για τις σχέσεις νότου-νότου. Εργαζόμαστε πάρα πολύ ενεργά, ειδικά στον τομέα του εμπορίου. Υπάρχουν πολύ περισσότερες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών και βεβαίω αυτό προωθεί και την ανάπτυξη. Η Task Force διαδραματίζουν ε, μεγάλο ρόλο σχέση με τα πολιτικά κόμματα. Το θέματος ε, όλης δουλειάς που έγινε με τα κόμματα στις ε, χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το έχουμε συμπεριλάβει στην Μίνιστρα Διάταξη. Προθούμε να ενδυναμώσουμε την ε, πολιτική κουλτούρα στην χώρα. Επίσης συνεργαζόμαστε με τα συνδικαλιστικές οργανώσεις που είπε ο κ. Σκοφού σε σχέση με την παρέμβαση της κυρίας Φλότρου. απουσιάζει αποχώρηση της αιθούσης. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γκάλερ. Ε, προφανώς ε, έχω υπόψη μου το έργο της αντιπροσωπείας σας, της αποστολής σας. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Γιωβάνη στο θέμα αυτό. Πρόκειται, δεν είναι θέμα αισιοδοξής ή απεσιοδοξής, απλά προσπαθούμε να συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε καθημερινά με τους πρωταγωνιστές τώρα σε σχέση με τα σχόλια του κυρίου Παντσέρη πρέπει να συνεργαστούμε με όλα τα κόμματα, όλους τους εμπλεκομένους. Όσοι πιστεύουν ότι οι χώρες αυτές οπισθοδρομούν, να πω το εξή, ότι τα Ισλαμικά κόμματα σε αυτές τις χώρες κάνουν, συνεργάζονται και συνασπίζονται με λαϊκά κόμματα. Κοσμικά. Τώρα ο πρέσβης Τέιλορ έχει το λόγο και του ζητώ να είναι σύντομος και λακωνικός ως Άγγλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συναλφός μου ο κύριος Λεόν ανέφερε πολλά ζητήματα οπότε μπορώ εγώ να αναφερθώ σε υποσύνολο αυτών. Αλλά αναφέρατε και θίξατε μερικά πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα να ξεκινήσω με τον κύριο Γκέιτς και άλλους που ρώτησαν ε, τι γίνεται με την συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ και ένα ερώτημα του κυρίου Τάνοκ νομίζω που ρώτησε το εάν θα συνεχίζαμε τη βοήθειά μας αν ε, η συνθήκη αυτή έπαβε να ισχύει το Κογκρέσο μας ανισχύει ε, όσο και εσείς και έχει θέσει έναν όρο σε όλη μας τη βοήθεια στην Αίγυπτο, στρατιωτική και μη. Ότι δηλαδή αυτή εξαρτάται από το να συνεχίσουν να τηρούν την συνθήκη ε, με το Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντικός όρος που έχουν θέσει. Εμείς ε, ως εκτελεστική εξουσία το παίρνουμε πολύ σοβαρά και ξέρω πως και οι Αιγύπτιοι το ίδιο κάνουν. Πολλοί από ε, ο κύριος Γκέιτς ε, ρώτησε επίσης για την, το πρόγραμμα της μουσουλμανικής αδελφότητας ως προς αυτό των αδελφών μουσουλμάνων. Ε, ξέρετε πως η ΕΠΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία περίοδο προεκλογική και αν δείτε και τα προγράμματα που ακούγονται ε, μπορεί και εκεί να παραπλανηθείτε. Δηλαδή υπάρχουν τα προγράμματα και μετά υπάρχει και η πολιτική που ακολουθείται όταν αναλάβει κάποιο την εξουσία. Δηλαδή είναι άλλο το πρόγραμμα και άλλο το τι γίνεται όταν κάποιο αναλάβει την εξουσία. Παρ' όλα αυτά εξετάζουμε και μας ενδιαφέρει το ποιες είναι οι προθέσεις και οι στόχοι και τα προγράμματα των διαφόρων μερών. Και γι' αυτό είμαστε σε επαφή μαζί τους. Ε, συζητούσαμε το εάν είναι σωστό να συζητάμε με Ισλαμικά κόμματα, Ισλαμιστικά κόμματα. Και η απάντηση είναι σαφώς ναι. ναι. Από το υψηλότερο επίπεδο. Και σκοπεύουμε να το κάνουμε τώρα για κάποια α, ε, πραγματάκια ε, Κύριε Μιλάν, δεν συζητήσαμε για την Αλγερία γιατί δεν αποτελεί μέρος τη ευθύνης ε, της δικής μου ή του κυρίου Λεόν. Ούτε η Συρία επίσης. Θα μπορούσε η Συρία εάν πάει προς μια δημοκρατική μετάβαση οπότε ε, θα μπορούσαμε να την στηρίξουμε αυτή τη χώρα όπως μπορούμε. Και την Ιεμένη επίσης. Το ερώτημα του κύριου Κοφόρντ για την κοινωνία των πολιτών. Πολύ σημαντικό και Οι διερμηνείς έληξαν την υπηρεσία τους γιατί δεν προειδοποιήθηκαν για τη δεκάλεπτη παράταση και γι' αυτό σταματάνε όλοι, όχι οι Έλληνες. Which will be, which are